Επιστρέφουμε στι απογευματινέ μα εργασίε που όπω βλέπω είναι πιο χαλαρέ από εκείνε του πρωινού. Το πρωινό είχε μεγάλη ένταση, πολλές, πολλή δουλειά είχαμε, ενώ τώρα θα είμαστε πιο ήρεμοι. Ξεκινάμε με το πρώτο σημείο της ημερησία διάταξη για το σημερινό απόγευμα σχετίζεται με την πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την πρόθεση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομία. Ο εισηγητή ε, δεν είναι παρόν και κυρία Μαρτσίνκετς, συγγνώμη, και θα αντικατασταθεί από την κυρία Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Έχει κάποια... Έχουμε κάποια υποχρέωση εδώ πέρα. Κοιτάξτε, παίζουμε σε αυτό το, στο μίνι τουρνό από το σφαίρο εκεί 5x5. Ήδη κερδίσαμε ένα παιχνίδι. Ελπίζουμε να κάνουμε και άλλε νίκε και να πάμε καλά σε αυτό το μίνι τουρνό. Τέλο πάντων, για τη σημερινή μα συζήτηση έχω να σα πω τα εξή. Ο κύριος Ματσινκέβιτς λοιπόν που έπρεπε να είχε μια υποχρέωση λοιπόν ε, ε έκανε αυτή την έκθεση όσον αφορά ε, το θέμα μας που έχουμε επομένω τους ε, οικονομικούς παράγοντες εκείνους οι οποίοι προσπαθούν να πετύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της επιχείρησης. Υπάρχουν εδώ διαφορετικοί τρόποι ε, διαφορετικές μάρκες, υπάρχουν ε, μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, ε, πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ακόμα και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό επίσης που είναι σημαντικό είναι το εξής. Τα κέρδη να χρησιμοποιούνται για σκοπούς κοινωνικούς. Και αυτό γίνεται με την παροχή κάποιων υπηρεσιών κοινού ενδιαφέροντος. Επίσης, βοηθούν τους μη προνομιούχους, αυτούς που έχουν ανάγκη σε κάθε κοινωνία. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Αυτούς που είναι περιθωριοποιημένοι για διαφορετικούς λόγους, ακόμα και λόγους υγείας. Τους βοηθούν να ξαναενταχθούν στην κοινωνία. Τους βοηθούν επίσης να βρουν κάποια δουλειά. Ε, ακόμα και τους ανάπηρους βοηθούν. Δεν μπορούν αυτοί να έχουν πρόσβαση παντού, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού στην αγορά εργασίας και με αυτόν τον τρόπο <clears throat> διευκολύνονται Είναι πάρα πολύ σωστή η πρωτοβουλία των κοινωνικών επιχειρήσεων. Είναι αξιόλογη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάνω σε αυτό το θεσμό. Θα πρέπει τώρα να αξιολογήσουμε το έργο αυτών των επιχειρήσεων. Θεωρούμε ότι βοηθούν την κοινωνία βοηθούν την ε, κοινωνική ένταξη των προσώπων που είπαμε, βοηθούν στην κοινωνική συνοχή. Αναμφίβολα θεωρούμε ότι βοηθούν και στην οικονομία κάθε χώρας. Γίνονται κάποιες επενδύσεις Υπάρχουν θέματα γραφειοκρατίας, υπάρχουν θέματα λογιστικά, τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Πρέπει να διευκολυνθούν αυτές οι επιχειρήσεις και θα πρέπει να μπορούν να χρηματοδοτηθούν όσο χρειάζεται. Αυτά προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα πολύ θετικά και θα βοηθήσουν. όσα προτείνει η Επιτροπή για τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς των επιχειρήσεων αυτών είναι πάρα πολύ σωστά θα και θα βοηθήσουν στο να γίνουν επενδύσεις πάνω σε αυτές τις εταιρείε. Υπάρχει επίσης μια θετική πρόταση όσον αφορά ε, τη δημιουργία ενός ταμείου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου. Ευρωπαϊκό. Πολύ σημαντικό. Μια που αυτές οι κοινωνικές επιχειρήσεις εκδίδουν μετοχές υπάρχει επομένως κάποιος σχετικός κίνδυνος αλλά το σημαντικό είναι η κοινωνική τους συμβολή άρα θα πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους από πολλές και διάφορες πηγές να κάνουμε επομένως ό,τι είναι δυνατόν ούτως ώστε να βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις όπως κάνουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. δεν είναι μεγάλε επιχειρήσει οι κοινωνικές επιχειρήσεις, δεν είναι τίποτα μεγάλα μονοπόλια. Ε, συνήθως είναι μόνο πρόσωπε ή διπρόσωπε εταιρείε και αντίστοιχα λίγε είναι και οι μετοχέ του. Δεν έχουν αναγνωριστεί όσο θα έπρεπε ακόμα και από τι τοπικέ κοινωνίε. Πολλές φορές γιατί απλώς ο κόσμος δεν ξέρει την ύπαρξή του. γιατί επίσης ε, κυριαρχούν κάποια στερεότυπα πολλές φορές ε, υπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις αντίον τους. Άρα αυτό που θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη είναι να αλλάξει η αντίληψη για αυτές τις εταιρείε. Άρα χρειάζεται κάποια ενημερωτική εκστρατεία. Να γίνει μια εκστρατεία παντού και όλοι οι Ευρωπαίοι να μάθουν περί τίνος πρόκειται. να μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις να τα καταφέρουν και να λάβουμε απόψη ότι έχουμε ένα τέτοιο 10% των επιχειρήσεων Ευρωπαϊκών που, που είναι τέτοιες ε, κοινωνικές επιχειρήσεις. Μιλούμε για 10.000 θέσεις εργασίας. Βλέπετε δηλαδή πόσο λίγες είναι και πόσες θέσεις απασχόλησης δημιουργούν. Επομένως θα πρέπει να βοηθήσουμε στο να εξελιχθούν, να προχωρήσουν. Χρειάζεται συνεργασία και έτσι να αξιοποιήσουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνουμε το λόγο στην σκιώδη Συγκίτρια Περιτρίτσια Τόγια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι με πολύ περήφανα μπορεί το Κοινοβούλιο να εξετάσει αυτή την πρωτοβουλία όπως και άλλες που έχουν έρθει ε, για τις οποίες, έχει, τις οποίες έχει ζητήσει η Κομισιόν, διότι αυτή η σειρά δραστηριοτήτων της Κομισιόν είναι απόρρια μιας έκθεσης που εγκρίθηκε στο Κοινοβούλιο για την Κοινωνική Οικονομία και περιλαμβάνε πολλές από αυτές τις προτάσεις και ζητούσε από την Κομισιόν να αναλάβει ισχυρή δράση υπέρ ε, οικονομικών φορέων της κοινωνικής οικονομίας διότι μιλούσαμε συνέχεια για κοινωνική οικονομία χωρίς τίποτα παραπάνω. Έτσι λοιπόν αυτό αποτελεί αποκύημα του των εργασιών του Κοινοβουλίου. Το γεγονός ότι η Κομισιόν δίνει μια σειρά από μηνύματα, στέλνει μια σειρά ε, μηνύματα, πρωτοβουλίες και έχει και το κοινωνικό ταμείο. Εμείς λοιπόν, για να συμπληρώσω όσα είπε η συνάδελφος, ε, με τα οποία συμφωνώ απολύτως, θα ήθελα να ζητήσω πιο έντονα ορισμένα πράγματα. Εδώ μιλάμε για πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες. Θα σας πω δύο-τρία σημεία που μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό να υπογραμμιστούν και τα οποία ωστόσο έχουν ήδη προβλεφθεί εν μέρη από τη συνάδελφό μας ε, που εκπροσωπεί την εισηγήτρια. Το πρώτο είναι το εξή γιατί η Επιτροπή για τη Βιομηχανία υποστηρίζει τέτοιες διατάξεις διότι α, σκοπός αυτός της έκθεσης ε, του Κοινοβουλίου ήταν ε, οικονομική φορείς ε, και πρέπει να υποστηρίξουμε την οικονομική τους υποκειμενικότητα σε αυτό το κοινωνικό τομέα ο οποίος δραστηριοποιείται με οικονομικούς όρους παρότι δεν πραγματοποιεί κέρδη. Θα πρέπει λοιπόν να τα ευνοήσουμε ακόμη περισσότερο αυτού του είδους επιχειρήσεις διότι στο επίκεντρο του δραστηριότητάς τους είναι να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ευημερία, όχι μόνο κέρδη. Μάλιστα καθόλου κέρδη. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό. Πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν αυτό το καθεστώς επιχείρησης για αυτές τις επιχειρήσεις. Σε αυτή την πρωτοβουλία υπάρχει ένας ορισμός που για τους ενδιαφερόμενους ε, φαίνεται σωστά διατυπωμένη η κοινωνική επιχείρηση, διότι είναι δύσκολο να ε, δώσουμε έναν ορισμό ο οποίος θα ταιριάζει για όλες τις χώρες, τις πολύ διαφορετικές χώρες μεταξύ τους. Αν αυτός λοιπόν ο ορισμός ε, είναι εντάξει όπως πιστεύω εγώ, ε, αν είναι εντάξει και κατά την άποψη των κοινωνικών επιχειρήσεων, θα μπορεί να διαβιβαστεί σε όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να υπάρχει σαφήνεια και να μην αλλάζουμε κάθε λίγο και λιγάκι. Το βλέπουμε και σε αυτό το προσχέδιο. Είναι σημαντικό το ζήτημα των οικονομικών πόρων που θα διατεθούν. Δηλαδή πρόσβαση στα χρηματοοικονομικά μέσα. Δεύτερον, και η κατάρτιση από την εμπειρία όλων μας έχουμε μάθει ότι πολύ συχνά υπάρχει καλή θέληση αλλά λείπουν τα χρήματα για την κατάρτιση των διαφόρων ε, επαγγελματιών. Η πρόσβαση λοιπόν σε υπηρεσίες εκπαίδευσης ε, θα βοηθήσει αυτούς τους ε, κοινωνικούς συνεταιρισμούς κατά κάποιο τρόπο να αποκτήσουν τις κατάλληλες ικανότητες. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι να τον ευνοήσουμε την κοινοτομία είναι σημαντική η ευνόηση της καινοτομίας. Πολλές φορές καλούνται οι διαφορεφορείς ε, και υπάρχουν ε, περιπτώσεις καινοτομίας όχι μόνο τεχνολογικής αλλά και διαχείρισης συμμετοχής. Πιστεύω ότι θα μπορούσαν να μάθουν πολλά στον κόσμο με πρακτικές αϊφόρες και στην κανονική οικονομία της αγοράς, διότι καινοτομούν και από αυτή την άποψη. Μάλιστα με την Ευρωπαϊκή Αρρωγή θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάποιο έργο πόλων ε, κοινωνικής διαχείρισης ε, που θα βελτίωνε την ποιότητα και σε άλλους τομείς. Τα διάφορα στερεότυπα μας κάνουν να θεωρούμε ότι μιλάμε για δραστηριότητες χαμηλού επίπεδου επαγγελματικού. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Εγώ έχω δει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις με ελλειπές προσωπικό και άποψη ικανοτήτων σε ορισμένες ε, υπορισμένες συνθήκες στις δικές μας περιοχές ε, παρέχουν και οικονομικές επιχειρήσεις ε, για παράδειγμα και οικονομικής υποστήριξης ε, σε εμά. δεν κάνουν δηλαδή μόνο δουλειές κυπουρικής χρειάζονται λοιπόν υποστήριξη χρειάζεται η δημιουργία καινοτόμων πόλων και τέλος υπάρχει το ζήτημα των δημοσίων συμβάσεων το τελευταίο σημείο που ήθελα να αναφέρω δεν λέω ότι θα πρέπει να ευνοηθούν στις δημόσιες συμβάσεις αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τίθενται σε μειονεκτούσα θέση η νομοθεσία για τις δημοσίες συμβάσεις ε, που προσέχει περισσότερο τις δαπάνες, το κόστος, ε, το, αναζητεί το χαμηλότερο κόστος, συχνά οδηγεί σε επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται το προσωπικό τους. Ενώ θα μπορούσαμε να ευνοήσουμε τέτοιου τύπου επιχειρήσεις που δεν μπορούν ε, να προσφέρουν το χαμηλότερο δυνατό κόστος και έτσι να αποφύγουμε πολλά προβλήματα. Πολύ λοιπόν θετική αυτή η πρωτοβουλία, πολύ θετική η δημιουργία νέων εργαλείων. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κάποια πράγματα στη δράση της Κομισιόν να είναι πραγματικά στοχευμένη και να βοηθήσει. Μιλάμε πολύ συχνά για την ανεργία. για τους άνω των 50 ετών και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει την επαγγελματική επανένταξη μορφές που, ανθρώπους που σε πιο ανταγωνιστικές αγορές δεν είναι πλέον δεκτές ε, ενώ σε αυτό το τύπο κοινωνικών επιχειρήσεων θα μπορούσαν να βρουν ε, μια επαγγελματική κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη συναδελφό Τόγια. Η κυρία Μπαρέα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πάρα πολύ σημαντική και παρουσιάζει ενδιαφέρον ακριβώς όπως ε, ε, είπαν οι συγκήτρια και οι σκιώδες και ε, είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι δραστηριότητες και αυτές οι επιχειρήσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι το διπλό αποτέλεσμα, διπλές εποπτήσεις που έχουν όσον αφορά το ότι πρόκειται τα κέρδη τους να ε, επενδυθούν στην ίδια την επιχείρηση αλλά και ο κοινωνικός του χαρακτήρας. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε το 10% επιχειρήσεων και μιλούμε για 11 εκατομμύρια, 11 εκατομμύρια μισθωτούς που εκεί εργάζονται. Οπότε θα πρέπει να ζητηθεί τελικά ε, το, το, κάτι να γίνει δηλαδή, γιατί ε, είναι ένας ολόκληρος κόσμος αυτές οι επιχειρήσεις και κανείς κανείς ζωή με αυτές. Οπότε θα πρέπει να ε, έχουμε εξοπιστία των πληροφοριών, ε, είναι κάτι το οποίο πρόκειται να ε, βελτιώσει την ε, έκδοση και διαχείριση των μετοχών τους ε, και βοηθάνε επίσης αυτές τις εταιρείε και στην κοινωνική συνοχή. Υπάρχει πάντως κάτι άλλο βασικό, αυτό το οποίο θέλω να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι εάν πρόκειται τελικά να έχουμε ένα ταμείο που να τις ενισχύει, θα πρέπει να μελετηθεί το ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτό το ταμείο και πώς πέραν των θεσμικών πώς μπορούν και μη θεσμικοί επενδυτές να, επενδυθούν, να, συγγνώμη, να ασχοληθούν και να αναφερθούν αυτό το ταμείο. Επίσης, είναι καινοτόμες επιχειρήσεις. Είναι επιχειρήσεις τις οποίες ε, τις τελεχών επαγγελματίες. Θα πρέπει να γίνει σχετική έρευνα για να μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε, για να είναι κερδοφόρες γιατί τη σήμερα ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο το οποίο επιτελούν και φυσικά και το ότι ε, δημιουργούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Θα ήθελα για όλα αυτά να μου απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας ευχαριστώ. Και εγώ εγκρίνω ένθρωμα αυτή την έκθεση. Την ευελιξία που αντιπροσωπεύει για το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν για πολύ καιρό θεωρούνταν οι κοινωνικές επιχειρήσεις βάρη. Οι επιχειρήσεις που επεβίωναν με τα βίας. Καταλαβαίνουμε ότι σήμερα σε μια σύγχρονη και πολιτισμένη οικονομία θα πρέπει να συνδυάσουμε τρεις τομείς. Έναν ιδιωτικό εμπορικό τομέα, έναν δημόσιο τομέα δημοσίων υπηρεσιών διαφοροποιημένο και υψηλής ποιότητας και έναν τρίτο τομέα κοινωνικής οικονομίας. Δηλαδή επιχειρήσεις με στόχο όχι την επιδίωξη του μέγιστου κέρδους αλλά με στόχο την ικανοποίηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών. Αυτός ο τρίτος τομέας των κοινωνικών επιχειρήσεων δεν περιορίζεται στις ε, φιλανθρωπικές επιχειρήσεις που οι, ούτε σε εκείνες που ε, επιχειρούν την επανένταξη των αναπήρων ή των ανέργων. Υπάρχουν επιχειρήσεις απολύτως φυσιολογικές που κινούνται από αυτή τη φιλοσοφία. Στη δική μου τη χώρα, στη Γαλλία, υπάρχουν επιχειρήσεις αμουβαίου ενδιαφέροντος, Μιτιουέλ, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τράπεζες που απασχολούν εξειδικευμένους εργαζομένους και συχνά υψηλά εξειδικευμένους και που είναι είτε συνεταιρισμοί, είτε αμοιβαίου συμφέροντο, είτε επιχειρήσει που δεν έχουν ως στόχο τη συσσόρευση κεφαλαίου ούτε την επιδίωξη του μέγιστου κέρδου. Μπορώ να σα αναφέρω μεγάλο πλήθο, ειδικότερα στο πλαίσιο των ε, ε, ασφαλιστικών εταιριών. Υπάρχει λοιπόν αυτή η λογική. Πολύ καλό λοιπόν θα ήταν να, την να τις αποκαταστήσουμε στη θέση που τους αρμόζει και να προωθηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να διασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους εν μέρη. Συμφωνώ με τις προτάσεις ε, που έγιναν για να πάμε λίγο πιο πέρα όσον αφορά τις πρωτοβουλίες, να τις επεκτείνουμε, αλλά θα ήθελα να χαιρετήσω αυτή την έκθεση και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε. Πιστεύω ότι μπορούμε να την τροποποιήσουμε κάπως ώστε να την κάνουμε ακόμη καλύτερη. Ευχαριστούμε. Κύριε Ήμπλερ. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, κυρία Νίμπλερ έχει το λόγο. Αν συγγνώμη, συμπαθάτε με. Πολύ κοντά καθόμαστε, οπότε δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Μία σύντομη παρατήρηση έχω. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω εδώ την γειτόνισά μου για την πολύ καλή παρουσίαση της γνωμοδότησης. Ε, μπορώ να ε, συμφωνήσω και με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Ε, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι η οικονομική υποστήριξη των ε, επιχειρήσεων ε, και μια ε, ε, σχετική οδηγία σε ευρωπαϊκό επίπεδο βοηθάει ε, τις επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι ε, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να είναι λίγο πιο προορατικό ε, όσον αφορά την συμμετοχή των επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, στους διαγωνισμούς δηλαδή που επιτρέπουν την επιχείρηση με την καλύτερη προσφορά να πάρει μια σύμβαση, αλλά κοινωνικές επιχειρήσεις ε, δεν μπορούν να είναι τόσο ανταγωνιστικές. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω όσον αφορά τις ε, δημόσιες συμβάσεις να υπάρχει προτίμηση. όχι απλά να μην είναι εις βάρος τους, αλλά να υπάρχει κάποιο πριμ, κάποιο ιδιαίτερο πλεονέκτημα. μια εκτίμηση μια θετική εκτίμηση των ε, προσφορών ε, των ε, κοινωνικών επιχειρήσεων. Ευχαρίστω θα υποβάλω σχετική τροποποίηση, τροπολογία και θα χαρώ αν την υποστηρίξουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη συνάδελφο Νίμπερ. Γκέρες Κορτίνες, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ήρθα γιατί ξέρετε, σήμερα ήμουν σε μια κρόαση για την κοινωνική οικονομία και ήρθε εγώ εδώ και σα συγχαρώ για το εγγραφό σα. Όμω, θα πρέπει να πούμε και δύο λόγια. Ότι για εμά του Ισπανού αυτού του είδου οι συνεργατικέ επιχειρήσει, αυτού του είδου οι συνεταιρισμοί είναι κάτι το θεαματικό από πλευρά εκπαιδευτική. Γιατί έτσι οι δαπάνε είναι πολύ λίγε. τα έξοδα είναι λίγα. Ε, έχει ωφελήσει πάρα πολύ τους ε, τους, τους, τους δάσκαλους γιατί μπορέσαμε έτσι να έχουμε ε, πολύ περισσότερα σχολεία γιατί 60% ε, περισσότερα σχολεία φτιάξαμε μια που όντας μέλη του συνεταιρισμού το συμπίνει οι δάσκαλοι, έτσι το σχολείο ήταν πιο οικονομικό και καλύτερο. Οπότε άρα αντίστοιχα θα πρέπει και εδώ να ενισχύσουμε την κοινωνική οικονομία γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι, ε, Ακριβώ το ίδιο κάνει και η Πορτογάλια όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματο υγεία. Κάνε κάποια κέντρα υγεία επί τη βάση, τη, βάση του, του συνεταιρισμού. Και έτσι δεν ήταν τόσο πολύ ή δεν ήταν καθόλου ε, κρατική επένδυση αυτά τα κέντρα υγεία. Α πούμε, ε, το ίδιο ε, μπορεί, θα έχει γίνει στι διοικητικέ μα ε, αυτόνομε περιφέρειες με του παιδικού σταθμού Επίσης, είναι δυνατόν έτσι να ελέγξει κανείς τι γίνεται με τα χρήματά τους, ε, τα έξοδα, επομένως δεν μπορούμε παρά να δώσουμε συγχαρητήρια ε, και σε αυτές τις πηγές αλλά και στην εισηγήτρια. Ευχαριστούμε κυρία Κούκοβιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα διερμηνία προς την γλώσσα μου τα σλοβενικά και είναι μια ευκαιρία τώρα να αναδείξουμε αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις και βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές σε κάθε χώρα και ε, είναι θέμα επιχειρηματικότητας των νέων γιατί πάρα πολλοί ε, και νέοι αλλά και λιγότεροι νέοι αγνοούν αυτόν τον θεσμό, αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Επομένως, θα πρέπει να δούμε, θα πρέπει να οργανώσουμε περισσότερες ακροάσεις να συμμετάσχουν εκείνοι οι οποίοι μετέχουν σε αυτές τις αξιόλογες πρακτικές αυτών των κλάδων. Θεωρώ ότι έτσι μας δίνεται μια αξιόλογη υπηρεσία για τέτοιες υπηρεσίες, γιατί στην Ευρώπη υστερούμε σε αυτόν τον τομέα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, έτσι μπορούμε να καινοτομήσουμε και να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε κάποιες ε, υπηρεσίες ε, υψηλής τεχνολογίας, πληροφορικής και για τους μεγαλύτερους που θα μπορούσε να καλύψει όλους αυτούς τους ε, ηλικιωμένους, ε, τους ε, κοινωνικούς επιχειρηματίες του ΣΥΠΗΝ. Όπως είδατε μπορώ να μιλήσω μπορώ να μιλήσω αγγλικά, αλλά θα ήθελα διερμηνία στα σλοβενικά. Σας ευχαριστούμε. Το, το λόγο τώρα έχει ο κύριος Χέλμα. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Όπως βλέπετε ε, πάρα πολύ στην Ευρώπη δεν, δεν ξέρουν ακριβώς τι θα πει ε, η κοινωνική επιχείρηση. Και εγώ σίγουρα το χέρι μου, ούτε εγώ δεν ήξερα ε, καλά καλά τι είναι. Όμως άκουσα τη συζήτηση και νιώθω περισσότερη σύγχυση. Κάποιος που έλαβε το λόγο είπε ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν βάσιμες ελπίδες να γίνονται αγωνιστικές και οπότε θα πρέπει να έχουν κρατικά δεκανίκια. Άλλος είπε για τέτοιες ε, ομάδες επιχειρήσεων ε, είπε ότι δημιουργούν κάποιες οικονομίες κλίμακος και άρα μπορούν να είναι ανταγωνιστικές. Τι γίνεται, αν είπε. Οπότε, τι, τελικά, τι κάνουμε, θέλουμε να επιδοτήσουμε κάποιους που το αξίζουν ή απλώς το κάνουμε ίσα ίσα για να δημιουργούμε τζίρο κάποια οικονομική δραστηριότητα. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα η Κομισιόν. Είναι εδώ ο κύριος Μπάλενς της Γενικής Διευθύνσης Αγοράς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα-πρώτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ε, ευχαριστήσει για ε, τα όσα είπατε οι περισσότεροι που κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με εμάς όσον αφορά αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα πρέπει να εξετάσουμε τη γνωμοδότησή σας στην Διεύθυνση Επιχείρησεων και Βιομηχανίας. Κάτι γνώμη μας, ο ρόλος και η θέση αυτών των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι ε, κάτι που ξεπερνά την ε, απλή φάση ε, της πάροχη των συγκεκριμένων υπηρεσιών στους ε, βάρους της κοινωνίας. Είναι ένα ατού, ένα χαρτί που βρίσκεται στα χέρια τη Ευρωπαϊκή οικονομίας. Και ε, βεβαίω οι επιχειρήσει αυτέ αποτελούν ένα πρότυπο οικονομικής δραστηριότητας ε, που είναι τελικά βιώσιμο, που είναι ανθεκτικό περισσότερο το παραδοσιακό και που είναι ότι πρέπει σε τέτοιου είδους καιρούς κρίσης και καιρούς μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι ε, τελικά βοηθά και την βιομηχανική πολιτική ε, μια τέτοια επιχείρηση σε σχέση με το ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τον βιομηχανικό μας ιστό. Για αυτούς τους λόγους με μια σειρά προτάσεων προτάσεις που ξεκίνησαν και με εκείνη την ε, πρωτοβουλία και τις άλλες προτάσεις μας που αναφέρθηκατε στη συζήτηση. Έχουμε επίσης και την πρόταση σχετικά με το Ταμείο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Έτσι θα τις βοηθήσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Επίσης έχουμε και την πρόταση της Επιτρόπης για μία αναθεώρηση των διατάξεων που διέπουν τις, ε, τις δημόσιες συμβάσεις. Επομένως έτσι θέλουμε να πλαισιώσουμε πέραν της οικονομικής πτυχής αυτές τις επιχειρήσεις. Θεωρούμε ότι βοηθούν για την επίτευξη όλων των στόχων για το 2020 για μια πιο εφόρο ανάπτυξη και πιο κοινωνική. Και τελικά είναι και πιο καινοτόμα αυτή η ανάπτυξη. Είναι η χαμή του δώρατος αυτής της επιχειρήσης για την πολιτική της καινοτομίας της κοινωνικής. Και όταν μιλούμε για κοινωνική καινοτομία εννοούμε καινοτομία σε όλη τη διαδικασία παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών και επίσης το, το, τα, κέρδη τελικά τα καρπώνει όλη η κοινωνία. Να λοιπόν πόσο βοηθούν την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης αυτής της Τώρα, όσον αφορά τα ερωτήματα ε, του, του τελευταίου, δεν θυμάμαι το, ποιος το είπε, να το πω στα αγγλικά, μια που στα αγγλικά υπευλήθηκε η ερώτηση. Θέλω να σας απαντήσω ότι βεβαίως και στην ε, Αγγλία, στην, στην Ευρώπη υπάρχει μια ποικιλία απόψεων σε σχέση με το τι θα πει κοινωνική επιχείρηση. Ποικιλία λοιπόν από χώρα σε χώρα, ποικιλία αντιλήψεων. Ακόμα και στον ίδιο αυτόν τον κλάδο έχουμε ποικιλία μορφών κοινωνικών επιχειρήσεων. Μερικές από αυτές έχουν και οδοσκοπικό χαρακτήρα, μερικές άλλες όχι. Μερικές από αυτές θα έπρεπε, θα μπορούσαν να έχουν την κρατική υποστήριξη. Αλλά όλο και περισσότερε από αυτές μπορούν να είναι αυτάρκες. Θα πρέπει να βοηθηθούν αυτές οι επιχειρήσεις, σε αυτή την προσπάθεια να σταθούν στα πόδια του. και πολλές από αυτές τις κοινωνικέ ε, επιχειρήσεις απομακρύνονται από την κουλτούρα της επιδότησης και πάνε προ τη, τη μορφή τη αυθεντικής επιχείρηση. Γιατί φυσικά πάρα πολλά νομικά πρόσωπα συγκροτούνται για να είναι επιλέξιμα για τέτοιες ε, επιδοτήσεις. Αυτό σημαίνει συχνά, αλλά πολλές φορές αυτές οι ίδιες εταιρείες, ακόμα και με τη σωματική μορφή, αποτελούν επιχειρήσεις όπω όπως το εννοούμε εδώ στην Ευρώπη. Οπότε αυτές έχουν να μας δείξουν το τι θα πει αηφόρος επιχείρηση. Γιατί εκεί αναπτύσσεται μια επιχειρηματικότητα στο επίπεδο τη διαχείριση, οπότε υπάρχουν και οι δυνατότητες που πρέπει να τι εκμεταλλευτούμε να γίνουν πρωταγωνιστές στην αγορά, να ανταγωνιστούν μέσα στην οικονομία. Γι' αυτό και σας λέω ότι δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της, ε, των διαφορετικών αυτών μορφών κοινωνικών επιχειρήσεων. Όλες αυτές μπορούν να είναι τμήμα του μελλοντικού επιχειρηματικού τοπίου στην Ευρώπη. Ό,τι ερωτήσεις ε, τυχόν έχετε, ευχαριστώ να απαντήσουμε. και να συζητήσουμε τι θα γίνει με τους ορισμούς, τι διαβήματα πρέπει να κάνουμε για να τις βοηθήσουμε, για την απασχόληση για τις επιχειρήσεις, για όλες τις συναρμόδιες ε, γενικές διευθύνσεις κομισιών. Ευχαριστώ να συνεργαστούν μαζί σας. Ευχαριστώ τώρα το λόγο για τα συμπεράσματα στην κυρία Χίπνερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που μίλησαν. Τους ευχαριστώ για τη συμβολή τους και για την πεποίθησή τους ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να βελτιωθεί, να διευρυνθεί. Ευχαριστώ τη συνάδελφο που επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ασχολείται διότι πράγματι μιλάμε για ένα επιχειρηματικό μοντέλο επιχειρηματικό σημαίνει ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε χρήματα για παράδειγμα και την κοινωνική ασφάλιση είναι μια επιχείρηση ουσιαστικά καταλαβαίνω ότι η Κομισιόν μας προτείνει να διευρύνουμε τον ορισμό ώστε να περιλαμβάνει όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας που συμπληρώνουν τα κλασικά μοντέλα, το βιομηχανικό και το εμπορικό μοντέλο που έχουν ως στόχο μόνο το κέρδος. Αυτό που υλοποιεί η κοινωνική επιχείρηση και που για εμάς είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι δημιουργεί θέσεις εργασίας παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός τεράστιου αποθέματος θέσεων εργασίας για τη βιομηχανία. Ε, μια άλλη ερώτηση που σημείωσα αφορά την αναγκαιότητα υποστήριξης φυσικά της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Αφενός μέσω επιχορηγήσεων, αφετέρου μέσω δανείων χαμηλού επιτοκίου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε και τις δύο κατευθύνσεις. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις ε, πολύ συχνά λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο. Εξού και η ανάγκη τους ε, να συνεργαστούν με τις τοπικές κοινότητες. Πρόκειται λοιπόν πραγματικά για επιχειρήσεις ε, εγκύτητας κατά κάποιο τρόπο. Όλες οι παρατηρήσεις που έκανα θα διαβιβαστούν στους συναδέλφους. Οι συνάδελφοι επίσης υπογράμμισαν την αναγκαιότητα δράσης για την κατάρτιση ατόμων τα οποία θα μπορούσαν να αφοσιωθούν στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Κάθε άτομο για το οποίο δημιουργείται μια θέση απασχόλησης ε, βοηθάει στην ε, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχουμε πολλές περιπτώσεις κοινωνικού αποκλεισμού στην Πολωνία ατόμων που ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας ε, και που δεν ήταν απαραίτητα περιθωριακοί. άτομο, που ωστόσο λόγω κάποιας ασθένειας ε, χρειάστηκε να εγκαταλείψουν το επαγγελμά τους και άρχισαν να αναζητούν μια άλλη επαγγελματική οδό. Είναι σημαντικό να βοηθήσουμε και αυτά τα άτομα στις, ε, στην επιδίωξή τους αυτή. Ωραία, ευχαριστούμε Τετάρτη, 31 Μαΐου δηλαδή, αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι, είναι η τελευταία προθεσμία για τις τροπολογίες. Ψηφοφορία έχει προβλεφθεί για την 19η Ιουνίου, 10 Ιουλίου ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόλησης και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια δεν έχει ακόμα οριστεί. Τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σημείο, Εράσμο για όλους, το πρόγραμμα της Ένωσης για την παιδεία, την επαγγελματική κατάρτιση, την νεολαία και τον αθλητισμό. Έχουμε ως ε, συγγήτρια την Σίλβια Αντριάννα Τικάου, στην οποία δίνω τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το πρόγραμμα Erasmus for All καλύπτει την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την νεολαία και τον αθλητισμό. Σκοπό έχει να προετοιμάσει όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς για διαβίωμαθηση. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει και συνεχίζει υπάρχοντα προγράμματα, το Erasmus Mundus, το Tempus, το Αντολίν και το Alpha καθώς και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανοποιημένες χώρες. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι ένωση όλων αυτών των προγραμμάτων σε ένα, η ενοποίηση τους δηλαδή σημαίνει απλοποίηση, σημαίνει κοινού κανόνες που εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη-μέλη και λιγότερη γραφειοκρατία. Το Κοινοβούλιο και ειδικότερα η Επιτροπή Ήτρα έχει ζητήσει για όλα τα προγράμματα το προϋπολογισμό για την περίοδο μέχρι το 2020 ύψους 17,2 ε, εκατομμυρία ευρώ εκ των οποίων το 65% θα ε, χρησιμοποιηθεί για την κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού ε, ένα άλλο για το 4% για την υποστήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων και 2% για διοικητικές δαπάνες 318 εκατομμύρια ευρώ για τις δραστηριότητες Ζαν Μονέ και 238 εκατομμύρια ευρώ για μέτρα στον τομέα του αθλητισμού. Εκτός αυτών παραπάνω, ένα ενδεικτικό ποσό 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ θα δεσμευτούν για διαφορά εξωτερικά μέσα για την προώθηση ε, της εξωτερικής διάστασης της ανώτατης εκπαίδευσης. Έκανα πολλές προτάσεις. Πρώτα απ' όλα εμείς υποστηρίζουμε την απλούστευση του προγράμματος αυτού και την ενοποίηση όλων των προαναφερθέντων προγραμμάτων σε ένα διότι αυτό σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία για τους δικαιούχους. Ανάμεσα στις τροπολογίες που έχω υποβάλει, μπορώ να αναφέρω τη συμπεριλήψη εδώ της βιομηχανικής πολιτικής, διότι η βιομηχανική πολιτική εξαρτάται από την έρευνα και την καινοτομία στην Ευρώπη η διασφάλιση της πρόσβασης σε αυτό το πράγμα για τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ειδικότερα τους NGO που εργάζονται με τους νέους σε όλους τους παραπάνω τομείς, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτό το πρόγραμμα για άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα με σωματικά, οικονομικά, γεωγραφικά, πολιτισμικά και ούτω καθεξής προβλήματα Έχουμε απαιτήσει επιλεξιμότητα για εγγύησεις δανείων για τους ε, ε, φοιτητέ μεταπτυχιακών από μία χώρα που συμμετέχει σε, που σπουδάζουν για διδακτορικό σε άλλη συμμετέχουσα χώρα. Έχω ζητήσει για τον ορισμό στο παράρτημα 1 του κανονισμού αντί για κατεξοδότηση πράξης των κριτηρίων απόδοσης που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 11 ζήτησα να αποκλειστεί από τα κριτήρια ε, κατανομής ε, ε, με διαχείριση από Εθνική Αρχή των Κονδυλίων για την υλοποίηση των μέτρων του άρθρου 6 που σχετίζονται με το κόστος διαβίωσης του κράτους μέλος. Διότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε διακρίσεις μεταξύ προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ανάλογα με το κράτος ε, διαμονής τους. Έχω ζητήσει διαφάνεια και ε, το από την Κομισιόν να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της πληροφορίες ε, για τους καθορισμένες εθνικές αρχές, προγράμματα και τις αιτήσεις χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Έχω επίσης ζητήσει συνεργασία μεταξύ Κομισιών και κρατών μελών για τον ορισμό των εθνικών αρχών που θα είναι αρμόδιες για τη διαχείριση του προγράμματος και αυτό να λάβει χώρα έως την 1η Ιανουαρίου 2014. Ουσιαστικά οι τροπολογίες ασχολούνται με το δικό μας τομέα δραστηριοτήτων. Ζήτησα... Ε, ζητώ από τους νέους επιχειρηματίες να υποφεληθούν αυτού του προγράμματος. Έχουμε υποβάλει τροπολογίες για τους νέους επιχειρηματίες. Έχω συμπεριλάβω τη βιομηχανική πολιτική μεταξύ των πολιτικών που σχετίζονται με αυτό το πρόγραμμα και προσδοκώ να ακούσω τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των συναδέλφων. Και για άλλη μια φορά υποστηρίζω την απλοποίηση και την ανοποίηση των κανόνων, διότι αυτό σημαίνει λιγότερη γραφειοκρατία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Φόρντ, παρακαλώ. Um, thank you very much and thank... Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την κυρία Τικάο, όπως συνήθως, για την ε, σκληρή δουλειά που κάνει. Έχω κάποιους ε, συλλογισμούς ε, σχετικά με το θέμα αυτό. Καταλαβαίνω ότι συχνά το να ταξιδεύει κανείς εκτός της περιφέρειάς του ε, του κράτους μέλους του για να μάθει ε, μπορεί να έχει σημαντικό όφελος ε, και σημαντικό είναι η σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και τις επαγγελματικές δεξιότητες. Έχω όμως την ανησυχία ότι ε, τώρα που έχουμε περιορισμένα χρήματα ε, στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, των κρατών μελών, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα παρέχουν τις δεξιότητες αυτές με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ως προς το κόστος και το όφελος. Ε, καταρχήν έχουμε εδώ σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού και πρέπει να γνωρίζουμε από πού προέρχονται αυτά. Γνωρίζω ότι το 40% του προϋπολογισμού αυτού δεν ε, έχει ε, διατεθεί για κάποια συγκεκριμένη τομεακή προτεραιότητα και μήπως θέλουμε να το σκεφτούμε αυτό περισσότερο. Ε, έχω ανησυχίες όσον αφορά την ισορροπία, διότι μόνο το 2% των χρημάτων θα πάει στην ε, εκπαίδευση ενηλίκων ε, και όσον αφορά τα δάνεια για τα διδακτορικά, ε, αυτά πώς επικαλύπτονται με τα προγράμματα ε, που έχουν αποδειχθεί ε, πολύτιμα. Ε, μήπως έχουμε εδώ επικάλυψη εργασιών ή πράγματι δημιουργούμε προστιθέμενη αξία. Στο πρόγραμμα Jean έχουμε προστιθέμενη αξία αν ο στόχος είναι να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Προτείνω οι άνθρωποι που ε, τείνουν να συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά ε, Μάλλον πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί ήδη είναι ενημερωμένοι σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στόχος είναι να ε, κινητοποιήσουμε τον κόσμο να ταξιδεύει εκτός του κράτους μέλους του. Μήπως λέει θα πρέπει να στραφεί σε άλλον ε, τομέα ε, το πρόγραμμα αυτό και να ασχολούμαστε με επαγγελματικές δεξιότητες, με επαγγελματική κατάρτιση. Η δυνατότητα να καλύπτουμε όχι μόνο την επίσημη ε, εκπαίδευση αλλά και την ανεπίσημη εκμάθηση προηγούμενα προγράμματα έχουν βοηθήσει να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να φροντίσουμε να μην δημιουργήσουμε εδώ κενό. Όσον αφορά τον αθλητισμό, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη διάθεση δημοσίου χρήματο ε, στον αθλητισμό, ε, ωστόσο πρέπει να διατίθεται στοχευμένα. Είχαμε στις Βρυξέλλες ε, δύο-τρεις αργίες στις Βρυξέλλες και Τετάρτη απόγευμα σε ε, εργάσιμη μέρα ε, έχουμε ε, αθλητική εκδήλωση έξω από το κοινοβούλιο. Αυτό, αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με κοινοτικό χρήμα και αν ναι, τι μήνυμα στέλνει αυτό. Να βεβαιωθούμε ότι αν θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε τον αθλητισμό, τα χρήματα αυτά να δαπανώνται εκεί που είναι περισσότερο απαραίτητα και να τα δαπανούμε με λογικό τρόπο. Ευχαριστούμε το λόγο στην κυρία Γκουτιέρης Κορτίνες. Ευχαριστώ πολύ. Βρίσκομαι λίγο σε αντιφατική θέση. Ευχαριστώ κυρία Τικάο για τις προσπάθειές σας. Μ' αρέσει αρκετά το πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό, αλλά δεν νιώθω ότι αντικατοπτρίζει σωστά και συμφωνώ εδώ με ε, την ε, έκθεση της Επιτροπής Επισουσίας ε, ε, δεν νομίζω ότι αντικατοπτρίζει ε, τα προγράμματα για τη διαβίω εκμάθηση κτλ. Το να τα συνδυάσουμε όλα αυτά ε, υπό το όνομα Έρασμος που είναι ένα πολύ φημισμένο όνομα νομίζω ότι είναι κρίμα διότι επιτέλους η Επιτροπή έκανε κάτι καλό και τώρα το καταστρέφει αλλάζοντας την ονομασία. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την αλλαγή της ονομασίας. Δεν θα ήθελα να εξαφανιστεί αυτό. Ε, ε, η Επιτροπή Πολιτισμού προτείνει να το ονομάσουμε διαβίω εκμάθηση. Ε, αλλά το, ενώ το πρόγραμμα Έρασμος στόχο είχε τις ανταλλαγές ανάμεσα στα πανεπιστήμια μας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Πολλοί νέοι που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα Erasmus μπορούν να το γράψουν αυτό στο βιογραφικό τους. Ε, και έτσι λοιπόν ε, έχουμε προστιθέμενη αξία σε οποιαδήποτε εκπαίδευση με το πρόγραμμα ανταλλαγών έρασμος. Αλλά για ε, κάθε νέο ε, φοιτητή που προσπαθεί να ανεξαρτητοποιηθεί ε, είναι πολύ ε, σημαντικό το να μαθαίνει ξένες γλώσσες, να έχει σωστή εκπαίδευση κτλ. Και αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε το πρόγραμμα Έρασμος. Εμένα με απασχολεί ότι το επίκεντρο εδώ είναι η νεολαία. Εάν κοιτάξετε την κατάσταση στην οικονομική κρίση αυτή τη στιγμή, έχουμε πολλού επαγγελματίε οι οποίοι θα πρέπει να επανεκπαιδευτούν για να βρουν δουλειά σε άλλον τομέα. Μιλάμε για μια κοινωνία η οποία γυράσκει και φοβάμαι ότι η διαβίω εκμάθηση δεν έχει οριστεί σωστά για να λάβει υπόψη της και τους πιο ε, ηλικιωμένους εργαζομένους που θα πρέπει να παραμείνουν στην αγορά εργασίας. όλα αυτά θα πρέπει να ξεκαθαριστούν. τώρα με ενημερώνουν ότι το έρασμος θα ε, έχει διαφορετικές ε, ονομασίες. Φυσικά θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, πώς μπορούμε να σώσουμε το όνομα του έρασμου, ε, να αποφύγουμε όμως να καλύπτει τα πάντα. Η Βίκη Φόρντ αναφέρθηκε ε, στην ε, βιομηχανία που συμπεριλαμβανόταν στο πρόγραμμα αυτό, τώρα όμως έχει εξαφανιστεί. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι επίτροποι που θέλουν να αλλάζουν τα, τις ονομασίες σε όλα τα πράγματα. Είχαμε το Λεωνάρντο, είχαμε τη διαβίω εκμάθηση. Πρόκειται για δύο προγράμματα τελείωσε διαφορετικά και φαίνεται τώρα ότι ε, όλα αυτά τα αναζωογονούμε με διαφορετική ονομασία. Ε, οι πολίτες μας λοιπόν τώρα μπορεί να γνώριζαν ένα πρόγραμμα, τώρα να ψάχνουν να το βρουν αλλά μην το βρίσκουν επειδή έχει αλλάξει όνομα. Ε, η συνθήκη μιλάει για προγράμματα πλαίσιο. Έχουμε το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ε, τώρα έχουμε το Horizon 2020, το οποίο ουσιαστικά είναι η ονομασία μιας αεροπορικής εταιρείας. Ε, και περιμένουμε τον κόσμο να ψηφίσει τα προγράμματα αυτά το 2014. Δεν γνωρίζουμε όμως καλά καλά που βρισκόμαστε. Θα πρέπει να το εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Το πρόγραμμα αυτό έχει εκπονηθεί πολύ καλά. συγχαρητήρια στην ομάδα που το εκπώνησε είναι πολύ ωραία τα θέματα αυτά, αλλά λείπει η διαβίω εκμάθηση. Ε, η επανεκπαίδευση για να μπορέσει να βρει κανεί σε μια ε, άλλη δουλειά και θα πρέπει να τα συμπεριλάβουμε αυτά σε σχετικό μέσο. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, έχουμε κάποια καθυστέρηση, Δεν περιμέναμε να έρθει η συγγήτρια λίγο και έτσι αναλώσαμε λίγο παραπάνω χρόνο. Ε, Επίτροπε, ο Επιτρόπο έχει ήδη, ήδη έρθει, θα μα περιμένει λιγάκι. Τζόνσον, παρακαλώ. Γιωάννσον, συγγνώμη. Ναι, κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρότασή σας εδώ. Έχω κάποια σύντομα σχόλια και θα σας τα συμπεριλάβω σε ε, τροπολογής ε, στην Επιτροπή Ήτρε πιστεύω πρέπει να τονίζουμε περισσότερο την εκπαίδευση των ενηλίκων διότι τα προγράμματα που συμπεριλαμβάνονται τώρα στο Erasmus for All ε, συμφωνώ να έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα Erasmus for All αλλά φοβάμαι ότι η εκπαίδευση των ενηλίκων θα χάσει και ήθελα να τονίσω τη σπουδαιότητά της Επίσης ήθελα να πω ότι η διαβίου μάθηση είναι η μία πτυχή της. Και η άλλη πτυχή είναι πολύ σημαντική, είναι η εκπαίδευση ενηλίκων. Τώρα τα, ποσά, τα μεγέθη για το έτος 2035 που αναφέρονται εδώ είναι σημαντικό να είναι ε, μάλλον, συγγνώμη, η ηλικία των 35 ετών πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ε, μεγαλύτερε ηλικίε αν θέλουμε να μιλάμε για ε, εκπαίδευση ενηλίκων. Επίση, κατά την άποψή μα, είναι σημαντικό η επαγγελματική κατάρτιση να αναφέρεται εδώ με πιο ισχυρό τρόπο. Μεγάλο κομμάτι τη βιομηχανία και των επιχειρήσεών μα είναι τώρα παγκοσμιοποιημένο. Έχουμε δηλαδή και ανθρώπους ε, που ε, οι άνθρωποι δηλαδή που έχουν παρακολουθήσει επαγγελματική κατάρταση μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό διότι μπορούν να ανταλλάξουν και να ενισχύσουν τη δύναμη της Ευρώπης. Ε, εγώ συμμετείχα στις εργασίες για το Horizon 2020 και την περασμένη πέμπτη άκουσα από μια επιτροπή εμπειρογνώμων γερμανική για την κοινοτομία. Τώρα ανησυχούν για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, διότι παρουσιάζουμε έλλειψη συμμετεχόντων. Δεν έχουμε αρκετούς ανθρώπους και έτσι αποδυναμώνουμε την έρευνα, την κοινοτομία και την υλοποίηση. Πιστεύω και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα όσον αφορά λοιπόν τις πολιτικές ε, επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη αναφέρονται στο πρόγραμμα αλλά θα πρέπει να τις τονίσουμε περισσότερο και να είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνουν πραγματικότητα. Αυτά ήθελα να τονίσω λίγο παραπάνω και τέλος ήθελα να πω ότι στην εκπαίδευση σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα, ειδικά στις βόρειες χώρες, έχουμε ένα σύστημα εθελοντικής και φιλελεύθερης εκπαίδευσης και εκπαίδευσης που σχετίζεται με συνδικάτα. Και πιστεύω αυτή η πτυχή της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής, επειδή μιλάμε για ευρωπαϊκή ανταλλαγή, θα μπορούσε να προσθεθεί είναι πολύ σημαντικό πιστεύω οι ε, υπεύθυνα άτομα σε περιφέρειες, σε τοπικές αρχές να εμπλέκονται περισσότερο στο πρόγραμμα Εράσμους. Αυτά είχα να πω σχόλια και θα επανέλθω με τροπολογίες. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των συντονιστών. Ωραία, ευχαριστούμε. Έχουν ολοκληρωθεί οι ομιλίες. Τώρα έχετε ε, ομιλίες των δύο λεπτών στην συνάδελφο Μπαρέα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δύο σχόλια μόνο εκ μέρους μου. Θεωρώ ότι το πρόγραμμα Εράσμους υπήρξε μία από τις καλύτερες πολιτικές που υλοποίησε ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επέτρεψε στους νέους μας να γίνουν πιο Ευρωπαίοι και αυτό είναι θεμελιώδη σημασία στοιχείο. Ωστόσο, όπως είπα, υπάρχουν δύο πτυχές που θα ήθελα να ε, διευκρινιστούν περισσότερο. Η σχέση με τα κράτη-μέλη, μεταξύ των κρατών μελών, ένας από τους στόχους του προγράμματος Εράσμους θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη της κατάρτισης και μείωση της εγκατάλειψης των σχολείων. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Ε, αυτή είναι μια ερώτηση που θέτω και στην Κομισιόν λαμβάνοντας υπόψη επίσης ε, την ε, αναζήτηση πρώτης εργασίας για τους ε, αποφύτους και τους νέους επιχειρηματίες θα έχουμε κάποιες δυνατότητες απασχόλησης για αυτά άτομα που μόλις έχουν τελειώσει την εκπαίδευσή τους αλλά δεν βλέπουν καμία προοπτική από άποψη εράσμους. Θα πρέπει πιστεύω, ότι, θα πρέπει πιστεύω να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτούς καθώς επίσης και με τους ενήλικες. Ε, στην πρώτη λοιπόν ωστόσο έρευνα θα πρέπει να μελετήσουμε τους νέους που βρίσκονται σε πολύ ψηλά ενεργείας ε, που φτάνουν σχεδόν στο 50% στην Ισπανία. Ε, κύριε συναρφετικά, για τα συμπεράσματα σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Για να απαντήσω στο όσα είπε η συναδελφός, ε, προσδοκώ να λάβω τις τροπολογίες και σας διαβεβαιώ ότι θα τις εξετάσω με, ανοιχτό μυαλό και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε. Ε, τελικά θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα καλύτερο κείμενο. Τώρα για όσα είπε η κυρία Φούλντ, εάν προσθέσουμε τα, ποσοστότα, τα ποσοστά αναχωρήσεις, θα δείτε ότι δεν είναι 40% που δεν έχει εκχωρηθεί. γίνεται πολύ καλά η χώριση του προϋπολογισμού. Στο άρθρο 5 περιλαμβάνεται στους συγκεκριμένους στόχους στο γράμμα Α μιλάμε για αυτό που είπε η κυρία Γκουτιέρες Κορτίνες για την εκπαίδευση ενηλίκων. Πιστεύω και εγώ ότι όντως το Εράσμους είναι γνωστό και εκτιμάται ιδιαίτερα παγκοσμίως. Υποστηρίζω λοιπόν τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή του προγράμματος αυτού με τη συμπερίληψη πολλών άλλων προγραμμάτων υπό την ονομασία Εράσμου, διότι Εράσμους σημαίνει αριστεία και θέλουμε να έχουμε αριστεία στην εκπαίδευση. Είναι σημαντικό να απλοποιήσουμε, να ευθυγραμμίσουμε κάπως τους κανόνες. Το πώς θα το ονομάσουμε δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά το Εράσμους αποτελεί σήμα αριστεία στην εκπαίδευση. Γι' αυτό έκανα αυτή την πρόταση ε, να, ε, να, προτα... να συμπεριληφθεί στην πρόταση τη Κομισιόν ε, να συμπεριληφθούν όλα τα άλλα στοιχεία, η διαβίω εκμάθηση και η εκπαίδευση ενηλίκων. Θα σταματήσω εδώ, Πρόεδρε, για να ολοκληρώσω, το μόνο, για να συμπεράνω μάλλον, το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι προσδοκώ να λάβω τις τροπολογίες που θα βελτιώσουν τις διατάξεις οι οποίες αναφέρονται στην επαγγελματική κατάρτιση και στη συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες. Αναφέρομαι σε άνθρωπα άνω των 35 ετών γεγονός το οποίο δεν σημαίνει ότι όσοι είναι μεγαλύτεροι των 55 δεν είναι σημαντικοί. Ήθελα απλά να δείξω το γεγονός ότι το Εράσμους δεν ε, απευθύνεται μόνο στις νέες γενιές αλλά σε όσους θέλουν να μάθουν ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στη μεταβαλλόμενη κοινωνία στην οποία ζούμε. Μιλώντας για θέσεις εργασίας, ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις ήδη υπάρχουσες διατάξεις. Φυσικά η νεότερη γενιά ε, πλήττεται χειρότερα από την ανεργία από άλλες κατηγορίες ατόμων το εράσμος ε, καταπολεμά τη γραφειοκρατία, ευθυγραμμίζει τους κανόνες και τώρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε την επιτυχή υλοποίηση. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ τη συνάδελφο Τικάου για μια τελευταία πληροφορία. Ήθελα να σας πω ότι οι τροπολογίες μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 3η 5 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε την κυρία Βασιλείου, Επίτροπο Εκπαιδεύσης και Πολιτισμού που βρίσκεται εδώ μαζί μας και που είχε την υπομονή να περιμένει. Λυπόμαστε για αυτή την καθυστέρηση, οφειλόταν στην πολύ ε, σημαντική συζήτηση και έντονη συζήτηση που είχαμε εδώ. Σήμερα έχουμε συζητήσει δύο ζητήματα τα οποία σχετίζονται άμεσα με το δικό σας τομέα και σας δίνουμε αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Είμαι ευγνώμων για τη δυνατότητα αυτή να συζητήσω μαζί σας ε, το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας ε, και Τεχνολογίας. Ξέρω ότι το EIT έχει οδηγήσει σε μια πολύ καλή και πλήρη συζήτηση ε, μεταξύ σα ε, και ιδιαίτερα μεταξύ των εισηγητών ε, και των σκιωδών εισηγητών για το Ορίζον 2020 και το EIT και νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι μπορούμε να έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση πάνω στην πρόταση της Επιτροπής για την ανάπτυξη του EIT. Πρόκειται για κρίσιμη στιγμή. Καλούμαστε να διαμορφώσουμε την μελλοντική πολιτική καινοτομία τη Ευρώπη. Αποφάσει που σύντομα θα ληφθούν από το Κοινοβούλιο αυτό και από ε, τα κράτη-μέλη θα έχουν ε, διαρκή αντίκτυπο στην ε, δυνατότητα της Ευρώπης ε, να αντιδράσει γρήγορα σε οικονομικέ και περιβαλλοντικές προκλήσεις ε, και να προσαρμοστεί επιτυχώ σε τεχνολογικέ και κοινωνικές αλλαγές. Συζητάμε το πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε τι κατάλληλε συνθήκε για την καινοτομία και την ανάπτυξη στην Ευρώπη και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την δυνατότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίσει το μέλλον. Η ευμαρία της ε, Ευρώπης εξαρτάται εν μέρη από το πώς θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή βλέπουμε ότι υπάρχει ορμή, μια ορμή τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να, να προωθηθούν ε, οι επενδύσεις ε, που οδηγούν σε ανάπτυξη. Πολλές ε, κυβερνήσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν πολιτικές καινοτομία και απασχόλησης των νέων και πολύ καλά κάνουν. Και πολλοί συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων εδώ στο Κοινοβούλιο ζητούν πιο σαφή και πιο ισχυρή δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να, για να προωθηθεί η ανάπτυξη και η καινοτομία. Με πιο ισχυρό EIT έχουμε Ευρωπαϊκό ε, Ινστιτούτο Τεχνολογίας έχουμε ένα ισχυρό εργαλείο ε, για να ε, μπορέσουμε πράγματι να αλλάξουμε τον τρόπο που εμείς οι Ευρωπαίοι προσεγγίζουμε την καινοτομία. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει την οτροπία, να έχουμε, μια, να έχουμε έναν πολιτισμό με περισσότερη επιχειρηματικότητα και με στενή συνεργασία των πανεπιστημίων. Είμαι πεπισμένη ότι με την ανάπτυξή του το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας θα μπορέσει να βοηθήσει την Ευρώπη να καταπολεμήσει την ε, ανεργία των νέων, ε, ενισχύοντα τη συνεργασία ανάμεσα σε επιχειρήσει και πανεπιστήμια και βοηθώντα ε, να δημιουργηθούν και να οριστούν οι θέσει απασχόληση του μέλλοντο. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογία, κατά την αρχική φάση ανάπτυξή του, ήταν ένα πείραμα προώθησης νέων προσεγγίσεων, πραγματοποίησης ε, των αρχών ε, του ε, τριγώνου της γνώσης και ε, της ενίσχυσης ε, του πυλώνα της εκπαίδευσης. Επίσης, ήταν ε, πείραμα διακυβέρνησης στον τομέα της καινοτομίας της Ευρώπης, χάρη στην ευελιξία και αυτονομία του, αλλά και χάρη στην σημαντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και την δημιουργία των, των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας και των κέντρων με τα οποία συνεργάζονταν αυτά. Και παρά τον περιορισμένο θα έλεγα πειραματικό προπολογισμό του ήταν επιτυχές ε, πείραμα. Μέχρι το τέλο τη χρονιά, ε, το EIT θα έχει δημιουργήσει 20 εκπαιδευτικά προγράμματα, πάνω από 1.000 φοιτητέ θα έχουν συμμετάσχει μέχρι το τέλο τη χρονιά. Οι 27 νέες επιχειρήσεις ε, αναμένεται να έχουν ξεκινήσει τις εργασίες τους μέχρι το τέλος της χρονιάς και 35 διπλώματα ε, αναμένεται να εγκριθούν, να καταχωρηθούν. Η επιτυχία αυτή ε, ε, επιβεβαιώνεται από τους ε, βασικούς ε, εταίρους του EIT, του, την βιομηχανία, τα πανεπιστήμια, τους φοιτητές και τους επιχειρηματίες, τους οποίους συνάντησα πρόσφατα στις επισκέψεις μου στο Χόλμη και στο Βερολίνο. Είμαι πεπισμένη περισσότερο από ποτέ ότι το EIT αποδειχνεί, ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε το λεγόμενο ευρωπαϊκό οξύμορο, όπου έχουμε εκπαίδευση, έχουμε εξαιρετική βάση έρευνας, έχουμε δυναμικές βιομηχανίες και παρόλα αυτά σπάνια καταφέρουν τις καινοτόμες ιδέες να τις μετατρέψουμε σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή απλά ε, αποτυγχάνουμε να τα διαθέσουμε στην αγορά με τρόπο εμπορικά βιώσιμο. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνολογίας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεχνολογίας έχει ε, γίνει μια ελκυστική πρόταση για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ευρώπης. Ε, ένα σαφές μήνυμα ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Εξίσου σημαντικό είναι ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογία προσεγγεί πολλέ ε, ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες είναι κορυφαίες στον τομέα του, αλλά είναι πολύ μικρές για να έχουν σημαντικό αντίκτυπο από μόνες τους. Ε, αυτό το γεγονό από μόνο του ε, αποτελεί σημαντικό συμβολή στην ευρωπαϊκή πολιτική καινοτομία. Επίσης, έχει καταφέρει να έχει καταφέρει να συνδυάσει ε, εθνικές επενδύσεις 5 εκατομμύρια ευρώ από το Grand Pound στη Γαλλία και 50 ε, ε, εκατομμύρια σε διάστημα πενταετίας από μια πρωτοβουλία στη Γερμανία για να σας αναφέρω δύο παραδείγματα μόνο κάτι που ευθυγραμμίζει καλύτερα τους ευρωπαϊκούς με τους εθνικούς στόχους κάτι το οποίο επιδιώκουμε. Κυρίες και κύριοι, ναι, επιτυχία ναι, μια πολύ καλή ιδέα, αλλά μέχρι στιγμής ε, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας ήταν ε, μόνο ένα περιορισμένο πείραμα. Ε, η πρόκληση μα τώρα είναι να εφαρμόσουμε το πρότυπο αυτό σε μεγαλύτερη κλίμακα, ώστε η καλή ιδέα να μπορέσει να έχει ε, βαθύτερο και ευρύτερο αντίκτυπο. Ε, γνωρίζω ότι είναι δύσκολη και ευαίσθητη φάση αυτή, όπου είναι πολύ δύσκολο να παραστρατήσουμε, ε, να παραπλανηθούμε από την υπερβολική φιλοδοξία μας, όπως είναι επίσης να φοβηθούμε και να μην τολμήσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Τελικά όμως, εάν θέλουμε να ε, οδηγηθούμε σε αλλαγέ όσον αφορά την καινοτομία στην Ευρώπη θα πρέπει να δείξουμε πολιτική φιλοδοξία και τόλμη. Η Κομισιόν έχει στείλει σαφέ μήνυμα στι προτάσει τη για το διάστημα μετά το 2013. Ενσωματώνοντας το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογία στο πρόγραμμα Horizon 2020 θέλουμε να θέσουμε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογία στο κέντρο ε, μιας ε, ισχυρή και συνεκτικής στρατηγική καινοτομία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προτείνουμε σημαντική ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας με προϋπολογισμό 3,19 δισεκατομμυρίων ευρώ και με τη δημιουργία έξι νέων ε, κέντρων ε, γνώσης και καινοτομίας. Το μήνυμα είναι σαφές. Εάν η Ευρώπη θέλει να δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης για όλους, τότε οι ε, επενδύσεις στην καινοτομία θα πρέπει να είναι μια από τις βασικές προτεραιότητες μας και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας αποτελεί ένα από τα καλύτερα μας εργαλεία για να πετύχουμε το στόχο αυτό. Του τους μήνε μήνες είχα συναντήσει με αρκετού από εσά για να συζητήσουμε το νομοθετικό πακέτο το οποίο προτείνουμε. Οι συναντήσει αυτέ επιβεβαίωσαν την πίστη μου ότι συμμεριζόμαστε μια κοινή, ένα κοινό όραμα σχετικά με το ρόλο τη καινοτομία στην οικονομία και την κοινωνία. Άκουσα προσεκτικά τι ανησυχίε σα και τι ιδέε σα και θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία αυτή να σα ευχαριστήσω και πάλι που μοιραστήκατε ε, μαζί μου τις ιδέες αυτές. Ε, περιμένω με ενδιαφέρον ε, τις τα σχέδια εκθέσεων των εισηγητών σας που από ό,τι καταλαβαίνω θα οριστικοποιηθούν αύριο. Θα τις μελετήσω προσεκτικά και ελπίζω να έχω τη δυνατότητα να τις συζητήσω μαζί σας πολύ σύντομα. Στο μεταξύ θα ήθελα να θίξω μια σειρά από πολιτικά θέματα ε, τα οποία, όπως επιβεβαίωσαν οι συζητήσεις μου μαζί σας, είναι ζωτική σημασίας εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε την επιτυχία αυτής της φάσης ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας. Ε, καταρχήν, ε, μια γενική παρατήρηση για τον προϋπολογισμό. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε ισχυρό συμφέρον να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να στηρίξουμε ένα φιλόδοξο προϋπολογισμό για το ορίζον 2020 ως ε, μέρος ε, της ε, στρατηγικής για να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την κοινοτομία στην Ευρώπη. Ο καθένας από εμά γνωρίζει τις δύσκολες διαπραγματεύσεις που μας περιμένουν. Πιο συγκεκριμένα όμως, ε, αν θέλουμε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας ε, να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο ευρωπαϊκό τοπίο καινοτομίας, τότε θα πρέπει να του δώσουμε τα μέσα ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο προϋπολογισμός που προτείνει η Κομισιόν ε, ακολουθεί μια προσεκτική ανάλυση του του, του μοντέλου του κύκλου ζωής ε, των ε, κέντρων ε, γνώσης και καινοτομίας και βασίζεται στις πραγματικές εμπειρίες των τριών κέντρων γνώσης και καινοτομίας που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είναι υπερβολικός ο προλογισμός αυτός εάν λάβουμε υπόψη μας τον στόχο μας. Ε, συμφωνούμε ότι είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε την καινοτομία, αλλά για να είναι πραγματική η αλλαγή που θέλουμε να πετύχουμε, θα πρέπει να ε, ε, να αντικατοπτρίζεται στις προτεραιότητές μας όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Ο, ο προπολογισμό που προτείνεται για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογία είναι μόλι 3,5% του συνολικού προπολογισμού του ορίζον 2020 και μόλις 20% του προϋπολογισμού που ε, προβλέπεται για, την, ε, για ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα. Η αύξηση είναι σημαντική, μόνο όμως επειδή ήταν τόσο χαμηλό το σημείο κίνησής μας. Ε, πρόκειτο για έναν προϋπολογισμό που στόχο είχε απλά να ξεκινήσουν τα πράγματα. Εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει σημαντικά στην άριστη έρευνα. Τώρα είναι σημαντικό ε, να ανταποκριθούμε στις ε, ε, επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αριστεία στον τομέα της καινοτομίας. Γνωρίζω ότι με κάθε ευρώ που ξοδεύουμε θα πρέπει να, η χρηματοδότηση να τη στοιχεί στα αποτελέσματα. Δεσμευόμαστε να έχουμε μεγαλύτερο και πιο διαφανή βαθμό λογοδοσίας που να ξεπερνάει αυτά που ισχύουν αυτή τη στιγμή ε, σε μέσα που σχετίζονται με την έρευνα. Θα παρακολουθούμε στενά και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και τα ΚΙΚΣ, τα Κέντρα ε, Γνώσης και ε, Καινοτομίας και με αυτή τη βάση σκοπεύουμε να κατανέμουμε το, την ετήσια χρηματοδότηση για τα ΚΙΚΣ. Επίσης, ε, προτείνουμε το EIT να αποτελεί αντικείμενο μιας ενδιάμεσης αναθεώρησης ε, και η δεύτερη ε, φάση της χρηματοδότηση να παρέχεται με βάση τα αποτελέσματα μιας ανεξάρτητη αξιολόγησης. Τρίτον, όσον αφορά τον αριθμό των κικς που θα ξεκινήσουν, ε, θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι ένας από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας είναι να ξεπεραστεί ε, ο παρόν κατακαιρματισμό ε, στο ευρωπαϊκό τοπίο καινοτομία. Για να το πετύχουμε αυτό, ο στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε μια κριτική μάζα δυναμικού στους τομείς που θα είναι στρατηγικοί για το μέλλον μας. Για να πετύχουμε αυτή την αποστολή, τα ΚΙΚΣ θα πρέπει να φτάσουν ένα μέγεθος το οποίο να διασφαλίζει ε, διαρθρωτική και μόνιμη ε, επιρροή ώστε να μπορούν να ε, ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν θα πρέπει να σκορπίσουμε υπερβολικά το δυναμικό μας. Η ανάπτυξη του EIT δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος του βασικού του στόχου, να πετύχει ταυτόχρονα αριστεία και κριτική μάζα. Η τέταρτη μου παρατήρηση αφορά το δυναμικό του EIT, τη δυνατότητά του να αποτελεί την εχμή για να απελευθερώσει το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καινοτομία ε, πέρα από τα παραδοσιακά κέντρα αριστείας που έχουμε. Υπάρχουν αναπτυσσόμενα, ξεχασμένα ή απλά άγνωστα κέντρα αριστείας παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ε, ε, επιχειρηματίες και οι καινοτόμοι του μέλλοντος ε, ζουν, εργάζονται και σπουδάζουν παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις ή στα πιο γνωστά πανεπιστήμια ή στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε η δουλειά του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και των ΚΙΚΣ να μπορέσει να διαδοθεί στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό έχουμε εκπονήσει στην, στο, στο θεματολόγιο στρατηγικής καινοτομίας ε, μια σειρά από πρωτοβουλίες. Να σας τονίσω τις ε, σημαντικότερες από αυτές. Έχουμε το Fellowship Scheme, το πρόγραμμα εταίρων. Έτσι θα μπορούν, με αυτό θα μπορούν ε, ικανά άτομα να συνεργάζονται εντό ενός ΚΙΚ. Ε, θα ε, δημιουργούνται όμω και πιο στενό σύνδεσμος ανάμεσα ε, στα ιδρύματα από τα οποία προέρχονται και τα κέντρα αριστείας που ανήκουν σε ένα ΚΙΚ. Έτσι, οι εμπειρίε και οι πρόοδοι που σημειώνει ένα ΚΙΚ θα αντικατοπτρίζονται και θα ενισχύονται σε άλλα κέντρα αριστείας σε όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα εδώ να ξεκαθαρίσω ένα σημαντικό σημείο. Τα ΚΙΚ δεν είναι κλειστά ε, κέντρα ε, σε τακτική βάση ε, ενσωματώνουν νέα μέλη είτε ως εταίρους είτε ως πλήρη μέλη. Και αυτό ήδη συμβαίνει στο εργαστήριο τεχνολογιών, στο εργαστήριο ICT στο Τρέντο ε, και αυτό είναι που κάνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας τόσο ελκυστικό. Η ευελιξία στην ε, διαχείριση ε, του δυναμικού ανάλογα με την ανάπτυξη των αναγκών του. Τέλος, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για τις συνέργειες. Η η φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε μια ισχυρή και συνεκτική στρατηγική καινοτομία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. η δομή του Horizon 2020 θα ενθαρρύνει συνέργειες ε, και συνεργασίες ανάμεσα σε όλα τα διάφορα ε, μέσα και σε όλες τις φάσεις του κύκλου ε, προγραμματισμού, ξεκινώντας από την επιλογή των ΚΙΚΣ ε, και ε, καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής και της διάδοσης των αποτελεσμάτων. Στον τροποποιημένο κανονισμό προτείνουμε ήδη κατά τη φάση επιλογής τα νέα ΚΙΚ να πρέπει να επιδεικνύουν την ετοιμότητά τους και τη δυνατότητά τους να δημιουργούν συνέργειες με άλλες πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνέργειες ήδη βλέπουμε στα τρία υπάρχοντα ΚΙΚ και έχουμε έτσι ένα αποτέλεσμα καταλήτη ή ένα αποτέλεσμα πολλαπλασιαστή το οποίο βρίσκεται στην καρδιά ε, του αντικτύπου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογία. Αυτό ακριβώ επιδιώκουμε. Πρωτού λοιπόν ε, κυρία Πρόεδρε σα ξαναδώσω το λόγο θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία να πω λίγα λόγια σχετικά με την πρότασή μα σχετικά με τι δράσει Marie Curie εντό του πλαισίου του Horizon 2020 διότι Ξέρω ότι πολλοί από εσέ ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το πρόγραμμα αυτό. Το πρόγραμμα ε, δράσης Marie Curie αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ε, δημιουργίας ε, της του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας με προϋπολογισμό ύψους 5,74 δισεκατομμύριων ευρώ για το προσεχές διάστημα που αντιπροσωπεύει αύξηση ύψους 21%. Ο στόχος παραμένει να στηρίξουμε την ανάπτυξη της ε, σταδιοδρομίας και την εκπαίδευση των ε, ερευνητών ε, με επίκεντρο στις δεξιότητες που σχετίζονται με την καινοτομία σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους με αύξηση της κινητικότητας. Προτείνουμε ένα νέο πρόγραμμα για ευρωπαϊκό διδακτορικό σε συγκεκριμένους τομείς διεύρυνση του προγράμματος ε, CoFund και απλοποίηση μια σειράς δράσεων. Ε, πρόκειται για προγράμματα τα οποία έχουν ε, αποδείξει την αξία τους, κυρίες και κύριοι. Αυτές ήταν οι εισαγωγές μου παρατηρήσεις και προσλέπω σε μια καλή συζήτηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, προς την κυρία Επίτροπο. Και Έχουμε μισό λεπτό, συγγνώμη 30 λεπτά για την ε, συζήτηση, οπότε και θα υπάρξει η δυνατότητα να λάβετε το λόγο και να ρωτήσετε και να απαντήσετε. Και πρώτα-πρώτα ξεκινούμε το λόγο στην κυρία Μαντουρέλη. Α, Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πίτροπε για την ευκαιρία που μας δίνετε να συζητήσουμε και πάλι μαζί σας όλα αυτά τα θέματα. Ε, αισθανόμαστε τυχερές ε, που έχουμε μπορέσει τόσες φορές να τα πούμε. Οπότε με την ευκαιρία που είστε εδώ θέλω να σας θέσω κάποια ερώτηση. Θέλω να σας πω πρώτα πρώτα ε, τις ανησυχίες που γνωρίζετε και τα, ε, από πλευράς δικής μου και από πλευράς ε, των συναδέλφων εδώ στην ε, Επιτροπή, την Κοινοβουλευτική αλλά και γενικότερα στην πολιτική μας ομάδα για αυτό το τόσο σημαντικό νομοθέτημα ε, και το σημαντικό αυτό ε, ίδρυμα της ε, καινοτομίας και της τεχνολογίας και συμφωνώ με τα περισσότερα τα οποία μας εξηγήσατε. Το θέμα είναι βέβαια τι γίνεται στην πράξη. Ότι όλα έχουν κάπως διαφορετική διάσταση και βεβαίως θεωρούμε όπως, όπως το, το, θεωρώ και εγώ και, και πολλοί από τους ανθρώπους εδώ ότι με μικρή πρικοδότηση αυτό το ίδρυμα ε, απέδωσε αποτελέσματα σημαντικά. Οπότε θα πρέπει να συνεχίσει ε, τη, τη, τη λειτουργία του και να έχει τη διάθεσή του αυτό το Ίδρυμα ό,τι χρειάζεται για να επιτελεί το έργο του. Τώρα, για πέστε μας. Σε σχέση το πρόγραμμα Horizon 2020, ε, χρειάζεται να υπάρχει συνεργασία για να προχωρήσουμε, αλλά και από πλευράς αυτού του Ινστιτούτου Πέστε μας, τι γίνεται όσον αφορά τις περικοπές που στα πλαίσια του Horizon 2020 ε, θα γίνουν. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, ε, σας λέω ότι μας, μας απασχολεί και θα πρέπει να συζητηθεί. Και όλους εμάς που μας απασχολούν αυτά τα θέματα μας προβληματίζει Οπότε, τι θα γίνει. Δεν θα πρέπει να δούμε το ότι κάποιοι συνάδελφοι έχουν κάποιε επιφυλάξει για το τι θα γίνει, αν θα αυξηθεί ή θα μειωθεί τελικά η πρικοδότηση. Δεν μπορείτε να μα εξηγήσετε τι θα γίνει. Πάντως σε σχέση με το Horizon 2020 όλες οι πολιτικές ομάδες συζητούμε ότι είναι ανεπαρκής η πρικοδότηση. Πρέπει να πείσουμε το Συμβούλιο και εσείς και εμείς ότι χρειαζόμαστε πιο μεγάλη προοικοδότηση. Βέβαια, εάν ε, ήταν όλα ρόδινα, θα είχαν λυθεί τα προβλήματά μας με τέτοιους κοινούς αγώνες. Τώρα κάτι άλλο το οποίο επίσης μας απασχολεί. Τι γίνεται όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την πληροφόρηση στα πλαίσια του Ινστιτούτου αυτού για τη σχέση με το ορίζον 2020. Μόνο εκεί, μόνο εκεί έχουμε μια τέτοια δουλειά ε, γνώσης όσον αφορά την έρευνα, όσον αφορά την γενοτομία, όσον αφορά τη, τη γνώση. Και όπως και εσείς μας εξηγήσατε, χρειάζεται περισσότερη συνεργασία ε, ίσως και ενοποίηση του Ιδρύματος με τις υποτροφίες ε, Μαρία Κιουρί. Τι λέτε. Φυσικά τι πρέπει να λάβουμε υπόψη. Αυτό θα σας πούνε και οι συνάδελφοι. Ότι τα πανεπιστήμια, η κατάρτιση, η γνώση δεν πλαισιώνεται αρκετά από το πρόγραμμα Horizon 2020. Και για τα Kicks βέβαια Υπάρχει το ερώτημα. Τι γίνεται σε σχέση με τις πρωτοβουλίε από μια μεριά και με τα ΚΙΚΣ από την άλλη. Το ΚΙΚ καλύπτει και θέματα πληροφόρησης, αλλά τα κοινά προγράμματα όχι. Τι λέτε, τι διάκριση μπορεί να γίνει. θα πρέπει να κάνουμε κάτι για την αριστεία και για την καινοτομία. Να βελτιωθεί η κατάσταση. Να διευρυνθεί η δραστηριότητά μας όσον αφορά την αριστεία. Γιατί με λίγα χρήματα έχουμε πολλούς ερευνητές και ερευνητικά κέντρα που μπορούν να φτάσουν στην αριστεία. και για την καινοτομία έχουμε ένα σημαντικό όργανο, τόσο ώστε να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας. Άρα θα πρέπει και εν προκειμένου να αναβαθμίσουμε τις προσπάθειές μας, ώστε να ελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις. Ε, πολλές φορές έγιναν κάποιες απόπειρες οι οποίες απέτυχαν. Τι γίνεται και τι γίνεται με τις επικαλύψεις που έχουμε πώς θα, θα, θα άρουμε τις επικαλύψεις μεταξύ των βραβείων ε, Μαρή Κιουρί και του Έρασμος για όλους. Τι γίνεται με τη χρηματοδότηση των κοινών διδακτορικών. Έχουμε και αυτά τα κοινά διδακτορικά στα πλαίσια του Έρασμος Μούντος και από την άλλη μεριά έχουμε και τις ε, υποτροφίες Κιουρί και θέλετε να τα ενοποιήσετε και να όλα να πάνε στο, σύστημα των υποτροφιών Κυρία. Και τα κοινά δεκτορικά υπάρχει μία, ένας φόβος ότι δεν θα γνωδοτούνται στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και Πρόεδρος. Κύριε Ματίας, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε ξανά που ήρθατε. Που ήρθατε και συζητούμε όλα αυτά τώρα. Με συμφωνούμε τα περισσότερα που αναφέρατε, αλλά συμφωνούμε και με τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν. Όπως είπε και η κυρία Ριέρα Μαντουρέλ, και εγώ θέλω να τονίσω το πόσο σημαντικό θεωρούμε το Horizon 2020 για τα θέματά μας. Χρειάζεται μια συνέργεια μεταξύ έργων, προγραμμάτων, πολιτικών, ούτως ώστε κάτι να γίνει και για την περίπτωση της έρευνας όμως. Δεν έχουμε και πολλές ευκαιρίες τελικά για να προχωρήσουμε στην Ευρώπη, στη έρευνα και τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συγκυρία, κρίσιμη. Θα πρέπει επομένως να επεξεργαστούμε την καλύτερη δυνατή πρόταση ώστε να προχωρήσουμε σε αυτά τα μέτωπα. Για το 2020 θα πρέπει να προβληματιστούμε για το μέλλον της Ευρώπης. Συμφωνώ με τις περισσότερες ανησυχίες σας, αλλά και με τις λύσεις που προτείνετε. Άλλωστε, αύριο θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης, το σχεδοκειμένο έχουμε συντάξει για την ε, έρευνα. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς το πρόγραμμα που είπατε θα γίνει ίδρυμα. Ναι, ίδρυμα να γίνει και να μην είναι απλώς ένα σύνολο από κίξ. Θα πρέπει επομένω να πρικοδοτηθεί αυτό το ίδρυμα έτσι ούτως ώστε να μπορεί να επιτελεί το έργο του και ίσως θα πρέπει να πούμε μερικά λόγια παραπάνω για το τι διαδικασίες προβλέπονται για την επιλογή των ΚΙΚΣ. Πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και θα πρέπει να θεωρήσουμε ως θεμέλιο αφιτηρία την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά χρειάζεται περισσότερη ευελιξία. Και αυτό γιατί όλα τα ΚΙΚΣ δεν είναι ίδια θα πρέπει να δούμε τι κατάτμιση υπάρχει, τι επικαλύψεις υπάρχουν. Και επίσης να είμαστε ευέλικτοι όσον αφορά τον λειτουργικό επιχειρησιακό ας πούμε χαρακτήρα των ΚΙΚΣ. Τώρα για κατάρτιση, εκπαίδευση, παιδεία. Είναι πάρα πολύ βασικά στοιχεία αυτά για τα ΚΙΚΣ. Μόνο αυτό έχουμε, ούτω ώστε με τόσο σωστό τρόπο να μπορούμε να συμπληρώσουμε το τρίγωνο της γνώσης. Παιδεία, έρευνα, ιδιωτικός τομέας. Η καινοτομία είναι κάτι που το χρειάζεται πάρα πολύ η Ευρώπη. Το πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να δώσουμε δουλειά στους νέους. Άρα είναι πολύ βασική υπόθεση η παιδεία και η κατάρτιση. Η κάθε χώρα βέβαια έχει διαφορετικά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα στην Ευρώπη υπάρχουν πολλά προβλήματα για την κατάρτιση και εκπαίδευση των αυριανών επιστημόνων. Σε κάποια κατημέλη κατάσταση όπως ξέρετε κύριε Επίτροπε, είναι δραματική. Ξέρετε τι γίνεται στην Πορτογαλία. Ξέρετε τι γίνεται όσον αφορά την εκπαίδευση και τις υποτροφίες. Αναβολές, καθυστερήσεις στις πληρωμές, όλα αυτά υποθηκεύουν, δυναμητίζουν, σαμποτάρουν το μέλλον της Ευρώπης. Και θα πρέπει επομένως να προσπαθήσουμε περισσότερο να αναβαθμίσουμε τις χρηματοδοτήσεις και πληκοδοτήσεις. Και όχι το αντίθετο. Για τις υποτροφίες, κύριε λοιπόν, μας είπατε και δικαιολογήσατε ότι θέλετε οι υποτροφίες αυτές να διατηρηθούν. Γιατί έτσι μέσω του συστήματος αυτού οι νέοι επιστήμονες βοηθούνται. Έτσι θα δημιουργήσουμε ένα σώμα νέων Ευρωπαίων επιστήμονων. Όμως, ό,τι και να γίνεται, δεν αρκούν οι υποτροφίες Μαρία Κυρία. Πεςτε μας τη γνώμη σας, μήπως μπορούμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών μέσα και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Τεχνολογίας είναι κατακλείδη. Αυτές οι δράσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και για την απασχόληση στην Ευρώπη και για την καινοτομία. Όλα αυτά θα προηγουμένω να τα συναρθρώσουμε για να πετύχουμε τους κοινού στόχους που έχουμε τάξει. Ζήτω συγγνώμη. Η συνάδελφος μίλησε λίγο περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Όταν λόγο έχει κυρία Κούτια Ρεσπαρτίνες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω δύο ώρες για τα θέματα αυτά, αλλά τελικά μου δίνετε ένα τριλεπτάκι. Και θέλω να σας πω ότι τελικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ότι η έρευνα πλησιάζει την παιδεία. Και πάλι πολύ σωστό είναι το ότι θέλουμε ποιότητα, θέλουμε αριστεία. Και θυμάμαι ότι κάποιο γνωστό που δούλευε στον ΟΣΑ μου είπε ότι τα τελευταία χρόνια η Κομισιόν έχει αλλάξει 100% την ε, πολιτική της παιδείας. Για να δούμε. Τι γίνεται όσον αφορά την παιδεία. Γιατί η εντύπωσή μου είναι ότι και για τα ΚΙΚ τα προγράμματα είναι λογικό να θέλουμε να βοηθήσουν την ε, βιομηχανία μας που είναι θέμα προτεραιότητας. Και όλο ένα και περισσότερο προσανατολίζεται η παιδεία προς ε, αυτό προς, προς την εφαρμογή, τη βιομηχανική του ζυπήν. Όμως θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε ε, φυσικά ανθρώπινους πόρους που να μπορούν να απορροφηθούν και να μπορούν και να απορροφήσουν και την νέα τεχνολογία και για το ορίζον 2020 αλλά και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Καινοτομίας και Τεχνολογίας ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί το τι θα γίνει με το θέμα της παιδείας. Όμως, άλλο είναι να ενημερώνουμε τους ερευνητέ, άλλο είναι να φτιάχνουμε ερευνητέ και άλλο είναι να έχουμε ένα πρόγραμμα που να εκμεταλλεύεται τα αποτελέσματα της έρευνας. Σαν τα παιδάκια κάνουμε. Ε, που, που θέλουμε να απορροφούν τη, την αριθμητική, που θέλουμε να δημορφώνουμε προσωπικότητα και αυτό θα πρέπει να καλυφθεί. Αλλά δεν το κάνουμε αυτό. Ενώ ξέρουμε τι θα πει δυνατότητα του ατόμου να μαθαίνει. Ε, είδατε πώς φτάσαμε να, να φτιάξουμε ακόμα και τη μοριακή φυσική, να προχωρήσουμε. Και τελικά τι θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε μία επιστήμη που να βοηθάει για το μέλλον, να μην κοιτάει προς τα πίσω. Να τι θέλουμε στα πλαίσια του Horizon 2020. Θα πρέπει τα ΚΙΚΣ να αφορούν αποκλειστικά στην ε, γνώση και την παιδεία. Εδώ, το θέλουμε αυτό να είναι εθνική αρμοδιότητα. Μα τότε θα πρέπει 50% τότε, αν δεν είναι εθνική αρμοδιότητα, να, αλλάξουν, να αλλάξει η ύλη των σχολείων. Κάτι άλλο τώρα. Το θέμα αυτό είναι το αυτού τη ενιαία σύλληψη για την γνώση. Ε, πρόκειται για την, ε, για την αριστεία. Η αριστεία. Ε, είναι θέμα πολιτισμού. Και με εκπλήσει το ότι υπάρχει τέτοια, τέτοια, τέτοιος μονοδιάστατος χαρακτήρας των, των ΚΙΚ. Πώς θα έχουμε μια πολιτική της πόλης αν δεν υπάρχει κάποιο είδου ευελιξία τόσο ώστε να μπορεί να αλλάξει και να προσαρμοστεί η στρατηγική. Γιατί είναι τόσο συγκεκριμένα τα σκικ που δεν υπάρχει συστημική, συστημικός προβληματισμός. Θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία να εντοπίσουμε την πολυπλοκότητα. Και να υπάρχει επομένω μέσω της ευελιξίας μία, ε, μία όσμωση μεταξύ των διαφορετικών. Ε, ε, όπως ας πούμε σε ένα κτίριο θα πρέπει κανείς να προβλέψει ε, όλες τις διαστάσεις, ξέρω εγώ, όχι μόνο έχει γκαράζ, αλλά πού μπαίνει το αυτοκίνητο, πώς κανείς φεύγει από τον γκαράζ, πάει στη, από τη σκάλα ή από τον ελκυστήρα, άρα επομένως Ας πούμε, θα πρέπει κανείς να προετοιμαστεί για να μπορεί να αποδεχτεί τον τουρισμό. Και έτσι φυσικά θα συμβάλλουμε στο να βελτιωθεί η κατάσταση της οικονομίας και να υπάρχει ευημερία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρος. Το λόγο έχει συνάδελφος Φόρντ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Την τελευταία φορά που μίλησα για το EIT, ορισμένα άτομα από το γραφείο σας ε, ήρθαν και μου είπαν ότι κάνω λάθος. Θα προσέχω λοιπόν σε αυτά που λέω. Το EIT είναι ένας νέος οργανισμός και ζητά σημαντική αύξηση του προπολογισμού. Αυτά τα χρήματα θα έρθουν από κάπου. Δηλαδή θα δοθούν λιγότερα χρήματα σε, στο ERC, στις κοινωνικές προκλήσεις, ε, στη ε, επίπεδα ε, βιομηχανικής ηγεσία του Horizon 2020. Διαφορετικά θα έπαιρνα περισσότερα χρήματα. Αυτό που θέλω λοιπόν να διασφαλίσω είναι ότι σε σχέση με αυτές τις άλλες πτυχές πραγματικά θα καταφέρετε να προσφέρετε την προστιθέμενη αξία στα προγράμματα πλαίσια πριν γίνει κάποια έκκληση γίνονται πολλές διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες ώστε να διαμορφωθεί η κλίση για υποβολή προσφορών και να είμαστε βέβαιοι ότι τα χρήματα θα πάνε εκεί όπου υπάρχουν εμπειρογνώμονες και όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Πώς μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το ίδιο θα συμβεί με διαφανή τρόπο με το EIT. Όταν είπα ε, τα χρήματα να αποφέρουν αξία, το γραφείο σας μου είπε είναι εύκολο γιατί έχουμε πάντα το match funding του 75% και αν έχουμε match funding ε, για τη βιομηχανία θα πρέπει να ε, παρέχουν την αξία. Αλλά ξέρω ότι στο πλαίσιο των kicks το match funding για τα ICT e είναι αρκετά εύκολο. Δεν θέλουν πολλοί άνθρωποι να, θέλουν πολλοί άνθρωποι να επενδύσουν σε αυτό. Είναι εύκολο να, μάνει, να βγάλει κανεί λεφτά, να βγάλει λεφτά για να βρει λεφτά για την υγεία, για την επιστημιστική ανάπτυξη είναι πολύ πιο δύσκολο. Αυτό το 75% λοιπόν, για τα κέξ μου φαίνεται αρκετά δύσκολο εμπόδιο σαν να συγκρίνουμε μήλα με πορτοκάλια και τώρα για το ζήτημα της προστιθέμενης αξίας λέτε ότι έχετε την ενδιάμεση ανασκόπηση αλλά αν αποφασιστεί σε αυτή την ανασκόπηση ότι δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία μπορούμε να σταματήσουμε αυτά τα προγράμματα διότι αυτό ξέρω ήταν πάντα δύσκολο στο παρελθόν και το ε, σημείο που με δυσκολεύει περισσότερο σε ένα ταξίδι μου στη Σκανδιναβία νωρίτερα φέτος ε, συνάντησε επιστήμονες από τέσσερις σκανδιναβικές χώρες το πανεπιστήμιο του ενός από αυτούς συμμετέχει στο ΚΙΚ και μας είπε ότι η εμπειρία του ότι αυτό το ΚΙΚ έχει τόσα πολλά χρήματα που δεν ξέρουν τι να τα κάνουν οι άλλοι συναδελφοί ε, θύμωσαν διότι ε, είπαν μακάρι να είχα εγώ ας πούμε τόσα χρήματα για τα ERC αφού ασχολούνταν με αυτά πώς είστε βέβαιοι αν δεν ξοδευτούν τα χρήματα στο EIT μπορούν να επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δαπανηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα ήθελα λοιπόν να είμαι βέβαιο ότι αυτά τα χρήματα που εκχωρούνται στα επιμερούς να μπορούν να επιστραφούν σε άλλους τομείς επιστημονικούς εάν μπορούν να ξοδευτούν καλύτερα κάπου αλλού. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Χέλμερ. Η ιδέα της ε, κυρίας Φόρντ ότι ε, οι δικαιούχοι της ε, Γενοδορής Ευρωπαϊκής Ένωσης από μόνοι τους ε, θα δώσουν πίσω τα χρήματα για άλλους στόχους, δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει. Εγώ ως βουλευτής έχω το προνόμιο να έρχομαι στην Επιτροπή να ακούω πράγματα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, για το οποίο ήξερα πολύ λίγα πριν, τώρα πάλι λίγα ξέρω. Από τους ε, ανθρώπους όμως, από του ψηφοφόρου μου στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο, τους οποίους ε, αντιπροσωπεύω, κανένας δεν το γνωρίζει. Ο αντίκτυπος λοιπόν του EIT είναι να προσπαθεί να καθορίζει την διδακτέα ύλη στα διάφορα πανεπιστήμια. Μπορεί αυτό να μην είναι αλήθεια, λόγω αυτό έχω ακούσει. Ακούσαμε πολλά για την αριστεία, χθε άκουγα για δίκτυα αριστείας. Σήμερα ακούμε για κέντρα αριστείας, αλλά σίγουρα ε, αριστεία είναι κάτι παραπάνω από το να ξοδεύουμε κάποια εκατομμύρια ευρώ και να γράφουμε κάποιες ωραίες εκθέσεις. Τι κάνουμε τελικά για να πετύχουμε την ε, αριστεία. Στην Ευρώπη έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλά πανεπιστήμια. Ε, το ξέρω αυτό επειδή και εγώ πήγα σε ένα από τα πολύ καλά πανεπιστήμια της Ευρώπης, στο Cambridge. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι τι κάνουμε εδώ το οποίο πιστεύουμε ότι προσθέτει ή ότι είναι απαραίτητο να αντικαταστήσει τα ε, πανεπιστημιακά ιδρύματα που ήδη έχουμε. Δεν είναι σαφές ε, τι ακριβώς προσπαθούμε να πετύχουμε. Ε, κυρία Πρόεδρε, ε, στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, πριν κάποιους μήνες ήθελα να διαπιστώσω τι είχαμε καταφέρει με 30 εκατομμύρια ευρώ Ήθελα λοιπόν να γνωρίζω πώς είχαμε εξοδεύσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ και κατάλαβα ότι ε, είχαμε αγγίξει, είχαμε φτάσει 3.000 ε, ε, πρόσωπα, λιγότερο από το 1% των ανέργων στην Ευρώπη. Δεν, κατάλαβα, δεν τους βρήκαμε δουλειά βέβαια, απλά τους επηρεάσαμε. λοιπόν κυρία Πρόεδρε, προσπαθούμε να δώσουμε την εικόνα ότι κάνουμε κάτι χρήσιμο. Εγώ θα ήθελα όμως να βεβαιωθώ ότι πράγματι έχουν αξία αυτά που κάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Πρόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Επιτρόπε. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομο και στη συνέχεια ενδεχομένως αν χρειαστεί να επανέλθουμε σε αυτό θα βρούμε και άλλη ευκαιρία. Είμαι πεπισμένος ότι η βιωσιμότητα του πολιτισμού μας μπορεί να επιτευχθεί μέσω από υλοποίησης που έχει πυλώνες βάσει της αξιοπρέπειας του ατόμου βασίζεται επίσης και στο κοινό καλό. Εμείς ε, βρισκόμαστε σε αυτόν τον πυλώνα. Πρέπει να επενδύσουμε στο άτομο διότι αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο το οποίο μπορούμε να σκεφτούμε όπως ε, ε, μιλήσαμε και νωρίτερα για επιχειρήσεις που λειτουργούν με κοινωνικούς σκοπούς. Το κοινό καλό μπορεί εξα, εξασφαλίζεται από αυτές τις επιχειρήσεις. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να υπογραμμίσουμε ότι πράγματι θα γίνουν οι απολύτως αναγκαίες επενδύσεις και ότι θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουν πραγματικά το αντικείμενο αυτό. Έτσι λοιπόν εγώ ενθαρρύνω την ε, Επιτροπή να προχωρήσει αλλά να είναι και πολύ αυστηρή όσον αφορά τα γενικά κριτήρια για αυτές τις δαπάνες έχοντας συνείδηση του γεγονότος ότι επενδύουμε στους βασικούς πυλώνες του πολιτισμού μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριος ε, Μπανίστερο. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να υπογραμμίσω τη σπουδαιότητα της πρότασης ε, της Κομπισιόν. Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, σίγουρα όχι λιγότερα. Ακούγοντας τι μας λέει ο ακαδημαϊκός κόσμος, τα οι διάφορες σχολές, οι επιχειρήσεις, τα σχολεία, θα μπορούσαμε ουσιαστικά να κάνουμε πολλά περισσότερα στο πλαίσιο της συνεργασίας σε σχέση με το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Σίγουρα είναι πολύ καλό που έχουμε επιλέξει αυτά τα κέντρα ε, καινοτομία και γνώσης. Ωστόσο η Ευρώπη θα πρέπει να αξιοποιήσει τη συνεργασία μεταξύ των διαφορών πυλώνων. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ε, εντατικοποιηθούν τα πράγματα διότι εκτός Ευρώπης, στην Ασία και ούτω καθεξής οι εξελίξεις ε, είναι ταχύτατες. Χρειάζεται λοιπόν να σημειώσουμε ότι επενδύονται πολλά εκτός Ευρώπης. Δημιουργούνται πράγματα, υπάρχει καινοτομία και αν δούμε αυτό που κάνουμε εμείς ε, με ένα κίκ από εδώ και ένα κίκ από εκεί, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. είμαι σύμφωνος ε, ουσιαστικά αυτό ήταν ο σκοπός, ε, να μπορέσουμε να βρούμε σημεία αριστείας, ε, τομεί αριστείας που μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ του. Πρότασή μου λοιπόν ποια είναι. Ευελιξία σίγουρα ναι. Εάν τα κέντρα γνώσης και καινοτομία μπορούσαν να είναι μεγαλύτερα, τόσο το καλύτερο, εάν μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά. Τώρα, όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, πρέπει να τα επανεντάξουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μιλάμε για 183 δισεκατομμύρια για αυτού του τύπου τις δραστηριότητες. Ένα κομμάτι από αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για δραστηριότητες αυτού του τύπου. Λέμε, ναι, είμαστε κέντρα αριστείας, είμαστε πανεπιστήμια που συνεργαζόμαστε, Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς πού βρίσκονται αυτά τα άτομα. Τώρα, λοιπόν, πρέπει πραγματικά να βρούμε τους καλύτερους εταίρους. Είναι σαν ένα τρίγωνο. Τα καλύτερα προγράμματα πρέπει να βρίσκονται στην κορυφή του τριγώνου. Και στη συνέχεια πρέπει αυτά να δείχνουν το δρόμο για την καινοτομία στην Ευρώπη, στους υπόλοιπους, μέσω της ασφάλειας, διασφάλισης της ποιότητας. Υποστηρίζω λοιπόν πολύ αυτή την έκθεση και όλες αυτές τις προτάσεις. Δεν υπάρχει λόγος να δαπανάμε περισσότερα σε σχέση με τα ΚΙΚ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ιωάννσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να κάνω μερικά σχόλια για αυτή τη συζήτηση για τα κέντρα γνώση και καινοτομία. Κάποιοι συναδελφοί μου έκαναν ορισμένε ερωτήσει, αλλά ήθελα να πω ότι όταν κάναμε την πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή για το Horizon, άκουσα το σχόλιο ότι μιλούσαμε για πολλά χρήματα που αύξαναν τον προϋπολογισμό της προφορικής και ότι για τα ΚΕΙΚ θα έπρεπε να το κοιτάξουμε λίγο καλύτερα. Τώρα στους συναδέλφους που το ρώτησαν θα έλεγα ότι εγώ είχα την ευκαιρία πριν από μερικές εβδομάδες να βρεθώ στη Στοκχόλμη, επισκεφτόμουν κάποια κέικ μαζί με την κυρία Καρβάλιο και την Επίτροπο. Το μήνυμα που λάβαμε ήταν ότι ότι το... ήταν αρμόδια άτομα σε παγκόσμιες εταιρείε και αυτό που είπα ήταν ότι, απάντηση, ότι η συνεργασία με τα ΚΙΚ και το τομέα της πληροφορικής ήταν πολύ χρήσιμη. Ανέφερα και κάποιες άλλες δραστηριότητες και προγράμματα που έχουμε στην έρευνα και μου είπαν αυτό είναι ένα από τα καλύτερα διότι είναι ευέλικτο και ανοιχτό και παρέχει δυνατότητες ε, στις βιομηχανικές ε, εταιρείες να συμμετέχουν. Ήθελα να δώσω λοιπόν και αυτή την προσέγγιση, διότι προσπάθησα, όπως σας είπα την πρώτη φορά που το συζητήσαμε, να μάθω περισσότερα για αυτό το θέμα των ΚΙΚ. Επίσης ε, λένε ότι ορισμένε φορές για να συμμετέχουν οι βιομηχανοί δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, είναι και θέμα της κοινότητας που συμμετέχει σε αυτή τη συνεργασία. Έτσι είχαμε το παράδειγμα του EIT και τον ΚΙΚ. Είναι μια πολύ καλή κοινότητα για να δουλεύει κανείς σε αυτήν. Ήθελα να σας δώσω δηλαδή αυτές τις πληροφορίες ότι αυτές οι εταιρείε έχουν άριστη εμπειρία από, μέσω πολλών συνεργασιών ερευνητικών μεταξύ πολλών προγραμμάτων. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι αξιοπρόσεκτες Αυτό πιστεύω τώρα. Είναι η μου ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με το EIT και με τα KICS. Αλλά η ερώτησή μου προς την Επίτροπο είναι επίσης εάν υπάρχει αυτό το όραμα τα όλα μπορούν να γίνουν καλύτερα φυσικά. Ήθελα να σχολιάσετε επίσης, ε, υπάρχουν επίσης ζητήσει ε, με τους εκπροσώπους των διαφορών επιχειρηματικών ενώσεων διότι πιστεύω ακόμη σήμερα είναι λίγο βορειοευρωπαϊκά τα ΚΙΚ. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτά τα κέντρα γνώσης και καινοτομία. Θα θέλαμε να έχουμε μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση σε αυτό το τομέα. Και αυτό θα πρέπει να συζητάμε τόσο στο Κοινοβούλιο αλλά και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήθελα να σας δώσω λοιπόν αυτές μου τις εντυπώσεις ότι ώστε να μάθουμε περισσότερα από τις υπάρχουσες ε, συμπράξεις. Ευχαριστούμε η συναδέλφος Μέρκης. Thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε για την εξαιρετική σας παρουσίαση. Πιστεύω πραγματικά ότι εσείς και η Επιτροπή ολόκληρη προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε πολλά ζητήματα με το EIT και την πρόταση. Το πρόβλημα είναι ότι αν προσπαθήσετε να τα επιλύσετε όλα, εν τέλει ίσως ε, να μην λύσετε τίποτα. Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται το EIT είναι σαν να είναι το καλύτερο εργαλείο. Για μένα αποτελεί ερωτηματικό. Εάν το είχατε παρουσιάσει με έναν τρόπο ότι εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο πείραμα, διότι περί αυτού πρόκειται. Συναρπαστικό πείραμα βέβαια, διότι κατά κάποιο τρόπο όλη η Ευρώπη ακόμα βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο πείραμα και αυτό που θέλετε να πείτε είναι ότι θέλουμε να μας πείτε ότι δεν είναι εδώ ε, πείδημα στο κενό. Το έχουμε προσπαθήσει σε πιλωτική φάση τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα που πρόκειται να το ξεκινήσουμε και να δούμε κατά πόσο πραγματικά επιπλέει, δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα επιπλέψει, αλλά ουσιαστικά η ερώτησή μου είναι θέλουμε να το ρισκάρουμε γιατί μιλάμε για μια τεράστια πρόκληση. Σας παρακαλώ μόνο μην το παρουσιάσετε σαν την απάντηση προς όλες μας τις προσευχές διότι θα επικριθείτε σκληρά. Μην ανησυχείτε κύριε Επίτροπε, εγώ θέλω να πλέψω μαζί σας. Θέλω να συμμετέχω σε αυτό το πείραμα. Το ζήτημα είναι ότι πιστεύω ότι ακόμα και σε πειράματα πρέπει να είμαστε σοφοί και να κάνουμε σοφές επιλογές. Το κατά πόσο λοιπόν πιστεύω ότι αυτό το πλοίο θα έχει τη δυνατότητα να επιπλέψει θα πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες και τις επιπτώσεις των υπαρχόντων EIT και να βελτιώσουμε τους μηχανισμούς παρακολούθησης, να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση και να μειώσουμε το διοικητικό φόρτο. Και πρέπει να πω ότι ευχαριστώ τους συζητητές για την άριστη συνεργασία τους σε αυτό το θέμα. Υποστηρίζω σε μεγάλο βαθμό την ιδέα μιας πιο ανταγωνιστικής κατανομής της χρηματοδότησης των ΚΙΚ. Όπως υπόθηκε, επίσης, ώστε και τα μικρότερα και τα συντομότερες διαρκές ΚΙΚ να μπορούν να υπάρχουν και να ευθυγραμμιστούν με το Horizon 2020, ειδικότερα με τον πυλώνα 2 και 3. Τώρα κάποια άλλα ανησυχητικά ζητήματα. Αυτό που βλέπουμε συνήθως είναι ότι όταν θέλουμε να καταπολεμήσουμε κάτι ε, δημιουργούμε μια συγκεκριμένη δομή, δηλαδή για την καταπολέμηση της φτώχειας, για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, για την κοινωνική κοινοτομία. Ε, η κοινωνική κοινοτομία είναι κάτι οριζόντιο, πρέπει να υπάρχει παντού, δημιουργία θέσεων εργασία ε, και τη σκάλα που θα μα οδηγήσει στην αριστεία. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε. Πόσα κικ θα είναι συμπληρωματικά με τα EIT. Βλέπω ότι τώρα κάποια παρουσιάζονται ήδη ως ΚΙΚ. Βλέπω ότι προγραμματίζεται ένα ΚΙΚ για τις πρώτες ύλες. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε πώς θα συμπεριλάβετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περισσότερο στα κέντρα γνώσης και καινοτομίας. Ευχαριστούμε κυρία Καρβάλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την παρουσίασή σας, ευχαριστώ και τους ε, εισηγητές και συνεισηγητέ ε, για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας. Δεν συμμετέχω στην εκπόνηση τη έκθεση, αλλά ε, με ενδιαφέρει το ε, ορίζον 2020 και στο πλαίσιο αυτό είχα συζητήσει με πολλούς ενδιαφερομένους και όταν μιλώ με τον σχετικό τομέα οι τομεί που συμβάλλουν περισσότερο στην ευρωπαϊκή οικονομία, οι τηλεπικοινωνίε, ε, τα αυτοκίνητα κλπ. Αν ρωτήσουμε λοιπόν αυτές τι επιχειρήσεις, ποιο είναι το μεγαλύτερο σας πρόβλημα αυτή τη στιγμή, θα εκπλαγείτε με την απάντηση, αλλά δεν έχουν αρκετό προσωπικό με την κατάλληλη εκπαίδευση για να αναπτυχθούν όσο θέλουν. Στην αεροναυτική είναι ε, πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό και στο Κοινοβούλιο είχαμε σχετική συζήτηση. Ταυτόχρονα έχουμε τόσο υψηλή ανεργία στην Ευρώπη μεταξύ των νέων. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για τα πανεπιστήμια ώστε να προσαρμοστούν και να έχουμε υψηλά εκπαιδευμένους ανθρώπους σε υψηλό επίπεδο ε, με δεκτορικά, ώστε να μπορούν να ε, καλύπτουν τις ανάγκες ε, του βιομηχανικού τομέα. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, νομίζω ότι τα ότι Εάν συνδυάσουμε την έρευνα και την καινοτομία ε, με στόχο την εκπαίδευση των ε, νέων, ώστε και να καλύψουν τις, ε, ομάδες, τις ανάγκες των μεγάλων πανεπιστημίων, αλλά συγγνώμη, των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά και για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις επιχειρήσεις τους. Νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο προς όφελος της ευρωπαϊκής κοινωνίας και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Λαμβάνοντας ε, λοιπόν ε, υπόψη μας αυτή την πτυχή, νομίζω ότι Νομίζω ότι αυτό είναι ο βασικός στόχος ε, του προγράμματος αυτού και αποτελεί το διαμάντι της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε στο βιομηχανικό τομέα και στην κοινωνία αυτό ακριβώς που χρειάζεται. Αυτό είναι ο στόχος μας, λαμβάνοντας υπόψη. Το μέγεθος ε, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας θα πρέπει να το χρηματοδοτήσουμε λοιπόν ανάλογα. Πολύ ευχαριστώ να συνεργαστώ μαζί σας αν είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Σύμβουλο Τεχνολογίας για την διεύρυνσή του. Ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής Εμπαρόσο ε, έχει αναφερθεί, το τόνισε αυτό. Ε, με, συνδεόταν το θέμα αυτό με το πρόγραμμα Λισαβόνα 2010 μια Ευρώπη δηλαδή η οποία να ε, είναι η πιο ανταγωνιστική και βασισμένη στην στη γνώση οικονομία του κόσμου. Ε, μια τέτοια οικονομία χρειάζεται και καθηγητές πανεπιστημίων ε, και νηπιαγωγούς. Θα πρέπει λοιπόν όχι μόνο να έχουμε περισσότερη έρευνα, αλλά τα αποτελέσματα των ερευνών να μπορούμε να τα φέρουμε στις κοινωνίες μας. Στα νηπιαγωγεία, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στα λύκια ε, και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, κύριε Επίτροπε, σας παρακαλώ ε, κατά την χρηματοδότηση του προγράμματος να τονιστεί το EIT να διαδώσει τις γνώσεις που έχουν που αποτελούν αποτέλεσμα των ε, προγραμμάτων που έχουμε χρηματοδοτήσει και τα αποτελέσματα αυτά να ε, εισρεύσουν στα εκπαιδευτικά μας ε, συστήματα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το καθήκον της εκπαίδευσης για να δημιουργήσουμε την κοινωνία βασισμένη στη γνώση, αυτό θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρό μας και αυτό θα πρέπει να αποτελεί επίκεντρο και κατά τη χρηματοδότηση του προγράμματος. Ευχαριστούμε. Τελευταία ομιλία ο συνάδελφος Λάνστορφ. Ευχαριστούμε την Επίτροπο. Το τεράστιο χαρτοφυλάκιο σας περιλαμβάνει και την πολυγλωσία. Και θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι αφορά τη βάση της πολυγλωσίας ή κλασικές γλώσσες για πολλές γενιές. οι κλασικές γλώσσες. Για πολλές γενιές ε, η κλασική γλωσσολογία και οι κλασικές γλώσσες, τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά, αποτελέσαν τη βάση των εκπαιδευτικών προγραμματών στα πανεπιστήμια. Σήμερα εξαφανίζονται σταδιακά ακόμη και στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία όπου χρησιμοποιούσαν τακτικά τα λατινικά Παρατηρούμε βαρβαρισμούς, χρησιμοποιούνται τα λατινικά με ιταλική προφόρα και πιστεύω τα λατινικά χρειάζονται προσοχή μας διότι αποτελούν κομμάτι της κοινή μας πολιτιστικής κληρονομιάς μαζί με τα αρχαία ελληνικά. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά τι ε, υποεξαφάνιση γλώσσε. γλώσσες. Υπάρχουν γλώσσες στην Ευρώπη που αντιπροσωπούν τεράστια πολιτιστική κληρονομιά με πολύ μικρό όμως αριθμό μιλητών. Ήθελα να αναφέρω τα γερμανοσερβικά, τα γίντις που εξαφανίζονται στην Ευρώπη. Και η ερώτησή μου προς εσάς, κυρία Επίτροπε, είναι τι μπορείτε να κάνετε ώστε να προστατεύσετε αυτές τις γλώσσες, αυτές που ε, κινδυνεύουν να χαθούν ή τις γλώσσες των μικρών μειονοτήτων. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ όλους σας ε, για αυτή την πολύ πλούσια συζήτηση και τα σχόλιά σας. Πρώτα απ' όλα κύριε Ράντσοφ θα ήθελα να έρθετε μια μέρα στο γραφείο μου και να κάνουμε μια καλή συζήτηση για τις υποεξαφάνιση γλώσσες και για τις αρχές γλώσσες για τις οποίες ε, και εγώ δείχνω τεράστια προτίμηση ώστε να... διότι το θέμα της συζήτησής μας σήμερα είναι πολύ διαφορετικό Ας κάνουμε λοιπόν αυτή τη συνάντηση μια φορά. Όσον αφορά το EIT, πιστεύω ότι πολλοί από εσάς έχετε θέσει το ερώτημα του επωνομαζόμενου υπερβολικού προϋπολογισμού. Θα σας πω λοιπόν ότι για αυτό το λόγο έχουμε αυτή την περίοδο πειραματισμού με πολύ χαμηλό προπολογισμό και είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσετε ότι 300 εκατομμύρια για τρία χρόνια δεν είναι πολλά χρήματα. Παρά αυτόν τον πολύ περιορισμένο προπολογισμό πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία του των όσων παρήγαγαν αυτά τα τρία κικ. Έχουμε φύλλα δεδομένων που έχω δώσει στους συζητητές αν οποιοδήποτε από εσά θέλει να λάβει αυτά τα fact sheets, παρακαλώ ενημερώστε με και θα σας τα στείλω. Ειλικρινά, εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια κλίμακα για την καινοτομία, πιστεύω ότι αυτό που προτείνουμε είναι πιθανώς λιγότερο από αυτό που θα ανέμενε κάποιος διότι είτε πρέπει να το κάνουμε σοβαρά και να ελπίζουμε για συγκεκριμένα αποτελέσματα ή να μην το κάνουμε καθόλου. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Κυρία Φόρντ, αν μπορείτε να μου δώσετε το όνομα του οργανισμού που σας είπε ότι έχουμε διαθέσιμα κονδύλια τα οποία δεν μπορούμε να τα ξοδέψουμε, παρακαλώ πείτε μου το διότι θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτά τα κονδύλια για να καλύψω τα κενά που έχουμε ήδη εμείς για το 2012 έχουμε κενό 53 εκατομμυρίων για το 2012 και είμαι βέβαιη ότι αυτό το ε, κενό θα αυξηθεί το 2013 διότι αυτό μπορούν να απορροφήσουν τα ΚΙΚ σήμερα που έχουν αναπτυχθεί και το τι μπορούμε εμείς να τους προσφέρουμε είναι πολύ διαφορετικό. Μας λείπουν 53 εκατομμύρια φέτος. Και επειδή θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα χρήματα που τους δίνουμε ξοδεύονται όπως πρέπει και με αποτέλεσμα, γι' αυτό το λόγο και όλες οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Horizon 2020 μακάρι να είχαν αυτό το σύστημα παρακολούθησης που ε, που υιοθετήσαμε εμείς για τα EIT. Έχουμε υιοθετήσει αυτό το σύστημα παρακολούθησης σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα, σε επίπεδο KIC, EIT, Horizon 2020 και για το Ευρώπη 2020. Σε αυτά τα τέσσερα επίπεδα δεν δίνουμε τα κονδύλια αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι ότι έχουν ε, συμμορφωθεί και έχουν επιτύχει τα όσα έχουν υποσχεθεί. Επίσης όταν μιλάμε για την ενδιάμεση αναθεώρηση μιλάμε σοβαρά πράγματα και ρώτησε κάποιο, αν ανακαλύψετε στην ενδιάμεση έκθεση ότι το ένα κικ δεν λειτουργεί καλά θα το σταματήσετε φυσικά και θα το σταματήσουμε δεν έχουμε κανένα δισταγμό διότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίζουμε να ξόδευουμε χρήματα σε κάτι που δεν είναι επιτυχές Όσον αφορά την ιδέα των ΚΙΚ και κάποιος ανέφερε ότι πρέπει να έχουμε ένα κεντρικό οργανισμό. Πιστεύω ότι ένας συνδυασμός μεταξύ του EIT ε, ιδιαίτερα ανεξάρτητου οργανισμού που διοργανώνει τη διαδικασία επιλογής των ΚΙΚ, συντονίζει το έργο των ΚΙΚ, διαδίδει τα καλύτερα μοντέλα διακυβέρνησης και χρηματοδότησης στα ΚΙΚ και από την άλλη έχουμε τα εξαιρετικά αυτόνομα ΚΙΚ, τα οποία καθορίζουν τη δική τους εσωτερική οργάνωση, τη δική τους σύνθεση, τη δικό τους πρόγραμμα και τις δικές τους μεθόδους εργασίας. Αυτός είναι ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός που μπορούμε να προσφέρουμε. Και πιστεύω ότι πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο για τον περιορισμένο χρόνο που το έχουμε δοκιμάσει λειτουργεί. Ζητώ συγγνώμη κυρία Μέρκος αν ακούστηκα ε, ε, κάπως πομπόδης. Δεν είπα ότι είναι το καλύτερο εργαλείο. Είπα ότι είναι ένα, ελπίζουμε ένα καλό εργαλείο και είμαι αισιόδοξη ότι αν του δώσουμε την υποστήριξη που χρειάζεται τότε θα το καταστήσουμε ακόμη πιο επιτυχημένο εργαλείο. Και φυσικά πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν και συμφωνώ μαζί σας. Αλλά φυσικά για να καταστήσουμε κάτι γνωστό πρέπει να ξοδέψουμε χρήματα σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης που ακριβώς αυτός είναι ο τύπος δραστηριοτήτων που θέλουμε και το έχουμε τώρα στον κανονισμό μας αυτό το 4,4% του προϋπολογισμού αφιερώνεται ειδικά για αυτές τις δραστηριότητες διότι θέλουμε τα κικ και θέλουμε την ιδέα του EIT να διαδοθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, σε όλες τις περιφέρειες. Ήδη για παράδειγμα έχουμε το κικ της Σιβηρίας που βρίσκεται στη Βαρκελόνη, κάπου γύρω από τη Βαρκελόνη, αλλά ήδη εξαπλώνεται. Εξαπλώνει τις δραστηριότητες του σε ολόκληρη την Ισπανία και στην Πορτογαλία. Το έχουμε λοιπόν ήδη. Επίσης με το πρόγραμμα Fellowship που προτείνουμε ε, το να έχουμε έναν εμπειρογνώμονα ο οποίος εργάζεται σε μη, ένα σχετικά άγνωστο κέντρο αριστείας, αυτός ή αυτή μπορεί να έρθει σε ένα ΚΙΚ ή σε ένα ε, κέντρο ε, σχετικό να προσφέρει, να δουλέψει εκεί και να επανέλθει στο ε, δικό του οργανισμό με γνώσεις νέες με τις οποίες ανεβάζει το επίπεδο. Και συμφωνώ με όλους τους είπατε ότι θέλουμε να επεκτείνουμε την έννοια του EIT σε μια πραγματικά πανευρωπαϊκή έννοια. Διότι μόνο σε τέτοια περίπτωση μπορεί το EIT να αποτελέσει ένα πραγματικά ανταγωνιστικό φορέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Διότι ειλικρινά, όταν ακούμε τους Κινέζους τι κάνουν για την καινοτομία, τι κάνουν για την επιχειρηματικότητα, με φοβίζει, με τρομάζει. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι αν επιλέξουμε να δώσουμε όθηση σε αυτού του τύπου στις δραστηριότητες θα πρέπει να το κάνουμε σοβαρά και να αφιερώσουμε χρήματα. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τίποτα. Ήδη τα ΚΙΚ και το EIT λειτουργούν πολύ καλά και με τις δράσεις Marie Curie. Το καλό με αυτό είναι ότι οι υποτροφίες που λαμβάνουν οι δικαιούχοι του Marie Curie συγχρηματοδοτούνται από τους εταίρους του EIT, από τις βιομηχανίες, τις τοπικές αρχές, τις περιφερειακές αρχές. Δημιουργούμε λοιπόν αυτό το τύπο συνεργειών, τις οποίες χρειαζόμαστε μεταξύ του EIT και των λοιπόν φορέων, διότι όλοι πρέπει να συνεργαστούμε μεταξύ μας πιστεύω. Κάποιος σας ρώτησε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών ε, πτυχίων που δίνουν διάφορα άλλα πανεπιστήμια και ιδρύματα από αυτό που κάνει το EIT. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Πρώτα απ' όλα παρέχει όπως και πολλά άλλα καλά πανεπιστήμια παρέχει σοβαρή υψηλής ποιότητας επιστημονική εκπαίδευση. Ωστόσο, σε συνδυασμό με στιβαρή εκπαίδευση επιχειρηματικότητας και καθοδήγηση και εκπαίδευση αποτελεί κομμάτι των προγραμμάτων μας. Έχουμε άτομα εκεί στα κέντρα ε, στα οποία εκπαιδεύουν τους νέους για το πώς να προσεγγίσουν τις βιομηχανίες, ε, πώς να βγουν στην αγορά σε αυτά τα collocation centers και να συστέγασης και να προωθήσουν την επιχειρηματικότητα. Αυτού του είδους την οτροπία χρειαζόμαστε για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη που είμαι βέβαιη όλοι επιθυμούμε. Υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα ξαναβρούμε την ευκαιρία και στο μέλλον να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ, για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστούμε εκ μέρους όλης της Επιτροπής στο επανειδέν.